Colleghi, procediamo all'audizione pubblica sul... Συνάδελφοι, περνάμε στην δημόσια ακρόαση σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις ε, ανεπίλητες ε, σειράξεις με ιδιαίτερη έμφαση στο Νότιο Κάφκος και την υπερνηστερία. Η σύραξη στην Γεωργία το, Αύγουστο 2008 οδήγησε τον Κάφκασο στην πρώτη θέση των ειδήσεων και είχαμε μετά την ε, κατάψη του πυρός αλλά και την ε, παρακολούθηση της ε, κατάστασης ε, οργής. Ε, κατάντησαν λοιπόν ε, αυτές οι εξελίξεις, αυτές οι λεγόμενες παγωμένες σειράξεις ή ανεπίλητες σειράξεις. σε μια ανακοίνωση του 2004 η Κομισιόν ανέφερε πως στην, Ευρωπαϊκή, στην γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να παραμείνει στην οικονομική και πολιτική μόνο ανάλυση της κατάστασης, αλλά να προβλέπει και να καταστέλει τις ε, κρίσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο δηλώθηκε και στην δήλωση της Πράγας το 2009. Οι εξελίξεις ε, πέρυσι, όπως η ανατολική γειτονία, η συνθήκη της Λισαβόνας, ε, διορισμός ε, του ΣΥΠΑ της εκπροσώπου σε εξωτερικά ζητήματα μας δείχνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει ρόλο σε αυτές τις ε, σειράξεις, ε, τις ανεπίλητες. Το ψήφισμα που βέσαμε να εγκρίνουμε σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τον Νότιο καύσκασο αποτελεί καρπό αυτού του προβληματισμού. Το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Κυριλόφου τονίζει την αναγκαιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια συνεπή και συνεκτική στρατηγική που θα συντονίζει τις δράσεις της στις χώρες να καταστήσει αποτελεσματικές δράσεις της αλλά και στοχευμένες και εστιασμένες στο στόχο. Η σημερινή ακρόαση θέλει να δώσει κινητρά στον συγητή κατά τον προσδιορισμό αυτής της στρατηγικής. Έχω λοιπόν την ευχαρίστηση να καλωσορίσω σήμερα το απόγευμα τους εμπειρογνώμονες μας την κυρία Σαμπίν Φίσερ, την κυρία Σαμπίν Φράιζερ και τον κύριο Τζόναθαν Κοέν. Καλώς ορίσατε. Μετά τις παρεμβάσεις σας θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Ευγέννη Κύριλοφ για να παρουσιάσει το σχέδιο έκτασης ε, σχετικά με τον, τον Νότιο Κάφκασο σας ευχαριστώ λοιπόν για την εδώ παρουσία σας και παρακαλώ να παραμείνετε στις αρχικές παρατηρήσεις μέσα στο πλαίσιο των 10 λεπτών προκειμένου να διεξαχθεί η επιθυμητή συζήτηση. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Okay, Thank you very much and also ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που με κάλεσε για την ακρόαση αυτή. Μου ζητήθηκε να εστιάσω στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση σειράξεων, αλλά μια και συζητάμε το θέμα του Νοτιού Καυκάσου, θα προτιμούσα να εστιάσω σήμερα στις ε, σειράξεις της θα βρείτε κάποια στοιχεία για την υπέρνηστερία στην ε, παρουσίαση PowerPoint που σας διαβιβάσαμε. Δεν θα εστιαστώ όμως αυτά στην παρουσίασή μου. Ούτε πρόκειται να εστιαστώ στα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχω μόνο 10 λεπτά στη διάθεσή μου και νομίζω ότι αυτό θα μας έπαιρνε πολύ παραπάνω χρόνο. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι η ανάμειξη του της Ένωσης ε, σε ανεπίλητες σειράξεις ε, υπό την ευρία έννοια αυξάνεται σταθερά τα τελευταία 7 χρόνια. Και τώρα θα ήθελα να κοιτάξουμε κυρίως τα επιτεύγματα ε, και τις αποτυχίες, αν θέλετε, της δράσης αυτής στον Αντιοκάυκασο. Κάφκασο. Καταρχάς, να πω δύο λόγια για το τι έχουμε πετύχει. Όπως είπα, η συμμετοχή της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί από το 2003, από το διορισμό ε, του εκπροσώπου της Ένωσης για τον Νότιο Κάφκασο και γενικά μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πετύχει να εμβαθύνει τις διμερείς της σχέσεις με τις τρεις δημοκρατίες του Νοτιού Καυκάσου και επειδή είναι περιορισμένη η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην σύραξη του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Η ανάλυση μας θα περιοριστεί αναγκαστικά στην Γεωργία. Και όπως ξέρετε, στη Γεωργία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερωθεί ως βασικός φορέας για την επίλυση των σειράξεων και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο να δοθεί ένα τέρμα στον πόλεμο τον Αύγουστο του 2008, έχει αναπτύξει διάφορα μέσα για να αποφύγει υπερτροκλιμάκωση. Δεν πρόκειται να σας παρουσιάσω ε, αυτή τη στιγμή τα μέσα, γιατί θα τα βρείτε και στην παρουσίαση PowerPoint. PowerPoint. Τώρα, ως προς τα αρνητικά στοιχεία. Θα πρέπει φυσικά να ομολογήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και άλλοι διεθνείς παράγοντε, δεν ήταν σε θέση να εμποδίσει το ξέσπασμα του πολέμου τον Αύγουστο του 2008, παρά την εντονότερη συμμετοχή των τελευταίων χρόνων και των έντονων διπλωματικών προσπαθειών στις αρχές του 2008. Η Ένωση επίσης δεν μπορούσε να ασκήσει πίεση στη Ρωσία για να συμμορφωθεί πλήρως με την Συμφωνία ανακοχής, ούτε μπόρεσε να αποτρέψει τη δημιουργία ενός νέου σταδοξικού στη γεωργία. Δεν υπάρχει πρόσβαση στην Απχαζία και οι συνομιλίες της Γενέβης είναι πολύ ασαφές πλαίσιο. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όλα τα υφιστάμενα μέσα λοιπόν δεν αποδείχτηκαν ε, αποτελεσματικά. Όπως σας είπα δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανάμειξη στον Αγκόρνο Καραμπάχ, άρα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε την πολιτική μας εκεί. Άρα για να συνοψίσουμε να πούμε ότι έχει αυξηθεί η ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία, αλλά παρόλα αυτά η κατάσταση παραμένει αρκετά ευαίσθητη και φυσικά ο πόλεμος του 2008 περιέπλεξε την κατάσταση περαιτέρω στην Γεωργία και αυτό ασφαλώς επηρεάζει και την ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, να περάσω στα εμπόδια σε ό,τι αφορά μια πιο επιτυχή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των σειράξεων στον Νότιο Κάφκασο. Εγώ θεωρώ ότι ουσιαστικά υπάρχουν τέσσερα διλήμματα, τέσσερα στοιχεία τα οποία υποσκάπτουν αν θέλετε την επιτυχία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Καταρχάς, υπάρχει το δίλημα μεταξύ μιας προσέγγισης ε, που θα έχει ως βάση την επίτευξη αποτελεσμάτων ή την εθνικοτική ε, ιστό της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζονται ιδιαίτερα σε οικονομική και πολιτική ε, ανάπτυξη για να επιληθούν οι σειράξεις και η ιδέα είναι ότι προκειμένου να, μεταμορφωθούν σε σταθερές δημοκρατίες και εύρυθμα λειτουργούσες αγορές οι χώρες αυτές θα χρειαστεί εμπιστοσύνη προκειμένου να ενσωματωθούν στην ε, περιφερειά τους, στην περιοχή τους και όλα αυτά αποτελούν την καλύτερη λύση για το μέλλον. Για κάποια περίοδο φαίνεται ότι στην Νότια Σωτία αυτή η προσέγγιση ήταν ε, πολλά υποσχόμενη όπου είχαν ανοίξει κάπως τα σύνορα, αν θέλετε, και τα όρια μεταξύ των εθνωτικών μειονοτήτων. Αλλά αν υπάρχει διαίρεση μεταξύ του κράτους και των αποσχεστικών ε, περιοχών όπως γίνεται στην Οσοτία και στον Αγκόρνο Καραμπάχ, η προσέγγιση αυτή δεν ε, υποστηρίζει την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης. Αντιθέτως, αφενός η οικονομική ενίσχυση μπορεί να εμβαθύνει το χάσμα μεταξύ των εθνοτικών κοινοτήτων και θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε και το εξής επειδή ούτε η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία ούτε η Ανατολική Εταιρική Σχέση προσφέρουν ε, μια προπτική ένταξη στη Γεωργία προκειμένου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιορισμένες δυνατότητες για την υποστήριξη των ε, εσωτερικών εξελίξεων, ούτε μπορεί να εφαρμόζει και να επιβάλλει όρους. Και προφανώς δεν μπορεί να ξεπεράσει την, το πολιτικό βάρος τρίτων χωρών, όπως η Ρωσία στη χώρα αυτή ή της Αρμενίας ε, στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Παρ' όλα αυτά, με την προσέγγιση της ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίμησε την εθνοτική πτυχή των ε, σειράξεων. Το επόμενο στοιχείο αφορά τις διμερείς σχέσεις έναντι της διαμεσολάβησης και της οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Όλες οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Νότιο Κάφκασο ε, λειτουργούν μέσω διμερών σχέσεων με τα εν λόγω κράτη. Και αυτό φυσικά περιορίζει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δρά ως μεσολαβητής ε, σε περιπτώσεις σειράξεων και αυτό το είδαμε και στην Γεωργία, όπου η κυβέρνηση Σακασβίλη μετά τον πόλεμο ζήτησε πιο έντονη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των σειράξεων ως τμήμα της προσπάθειάς του για την ένταξη των ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Και αυτό συνοδεύτηκε από μια εθνικιστική έκκληση σε ό,τι αφορά τις περιοχές της απόσχησης. Και γενικώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε αντιληπτή ως σύμμαχος της γεωργιανής ε, κυβέρνησης από τις αρχές στην Απχαζία, το οποίο φυσικά περιόρισε τη δυνατότητά της να δράσει ως ουδέτερος διαμεσολαβητής. Σε ό,τι αφορά τον Αγκόρνο Καραμπάχ, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μεταξύ σκύλα και χάριβδης. Γιατί στο πλαίσιο του ENP και του EAP σκοπεύει να αναπτύξει σχέσεις, εταιρική ε, σχέσεις με την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Το γεγονός ότι αυτές βρίσκονται σε ε, ουσιαστικά για τον Αγκόρνο Καραμπάχ δυσκολεύει την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρίτο στοιχείο αφορά, σε ό,τι αφορά τις ε, αντιλήψεις και τις προσδοκίες των χωρών που πλήττονται από τις σειράξεις. Είναι δύσκολο πιστεύω, είναι μάλλον σημαντικό πιστεύω στην παρούσα φάση να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά αντιδράει στις ε, εξελίξεις και στις, ε, στα περιστατικά δεν δρά εκ των προτέρων προληπτικά και εδώ πέρα υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της σύραξη στη Γεωργία και στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Όπως είπα, προς τη Γεωργία έχει ανοίξει την πόρτα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ούτε η Αρμενία ούτε το Αγκόρνο Καραμπάχ δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αρμενία, επειδή είναι, η Αρμενία επειδή είναι αρκετά πλεονεκτική η παρούσα θέση της και το Αζερμπαϊτζάν. Επειδή επικρατεί ο φόβος ότι η πιο έντονη συμμετοχή της Ένωσης και η μεγαλύτερη διάδραση μεταξύ των εκπροσώπων της Ένωσης και των τοπικών αρχών στον Αγκόρνο Καραμπάχ θα μπορούσαν να δώσουν μια διεθνή νομιμότητα στην περιοχή, η οποία εν τέλει θα αποβεί εις βάρος του Αζερμπαϊτζάν. Και γενικά μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μεγαλύτερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό πηγάζει και από την γενικότερη νοοτροπία και αντίληψη περί διεθνών σειράξεων στην περιοχή που επηρεάζονται από γεωπολιτικές πτυχές οι οποίες δεν ε, συνάδουν αν θέλετε με τον τρόπο που η Ευρώπη ε, περιγράφει τον εαυτό της σε ό,τι αφορά δηλαδή τα περί ήπιας δύναμης. Άρα υπάρχει εδώ πέρα μια συνέπεια. Τελευταίο στοιχείο που ήθελα να αναφέρω είναι η έλλειψη συνεκτικής ε, στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα στοιχεία που ανέφερα θεωρώ ότι καταδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμα ε, μια ενιαία στρατηγική για την αντιμετώπιση των σειράξεων στην περιοχή. Και αυτό οφείλεται σε τρία αιτία. Καταρχά, επειδή η συνεργασία στην περιοχή δεν είναι πάντα όμαλη και η γεωργία, στην οποία έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί φορεί της Ευρωπαϊκή Ένωση, το καταδεικνύει αυτό κατεξοχήν. Κατά δεύτερον, υπάρχει διχασμός μεταξύ των κρατών μελών για το πού θα πρέπει να τεθούν οι προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής στον Νότο ή στον Βορρά και τρίτον, επειδή υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των κρατών μελών για θέματα που θα πρεπει να δεθουν οι προτεραιοτητες της ευρωπαικης πολιτικης στον νοτο η στον βορρα και τριτον επειδη υπαρχει μεγαλο χασμα μεταξυ των κρατων μελων για θεματα που αφορουν τις σχέσεις με τη Ρωσία. Και πάλι αυτό κατέστη ιδιαίτερα σαφές στην περίπτωση της Γεωργίας, γιατί οι δύο σειράξεις τα τελευταία χρόνια καταλήξαν σε άμεση σύγκρουση Γεωργίας και Ρωσίας, το οποίο παρέλυσε ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν της επέτρεψε να αναλάβει δράση παρά μόνο μετά τον πόλεμο. Βάσει της ανάλυσης λοιπόν αυτής, θα ήθελα να καταλήξω σε τρία συμπεράσματα, να αναφέρω τρία στοιχεία για το μέλλον της ε, μελλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής σε ό,τι αφορά την περιοχή αυτή και την επίλυση των σειράξεων. Θα πρέπει νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει την προσέγγιση της σε ό,τι αφορά την ε, επίτευξη αποτελεσμάτων και το να ακολουθούνται οι εξελίξεις. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να μην, να μην επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και θα πρέπει η πολιτική της Ένωσης να λαμβάνει υπόψη τις εθνοπολιτικές διαστάσεις, τις διαστάσεις ως προς την ταυτότητα που εμπλέκονται στις σειράξεις και αυτά να εμπλακούν ως στοιχεία στην ανάπτυξη της πολιτικής της. Κατά δεύτερον, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τα όρια των διμερών προσεγγίσεων επειδή είναι ευρύ και θεμητό το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής, θα πρόκειται μάλλον για ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα, αλλά θα πρέπει και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νομίζω ότι ο Τζον θα μιλήσει για την κοινωνία των πολιτών μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Να αναφέρω στο σημείο αυτό, επειδή είναι σημαντικό για τα δύο πρώτα στοιχεία, ότι για παράδειγμα η ιδέα της δέσμευσης χωρίς αναγνώριση αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Και νομίζω ότι θα πρέπει να τύχει υποστήριξης από την Ένωση. Τρίτον, Νομίζω ότι στη διαδικασία εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εναρμόνιση των διάφορων μέσων που συμμετέχουν στον Νότιο Κάφκασο, καλύτερη συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής, με την ύπαρτη εκπρόσωπο και την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Όλα αυτά είναι πολλά υποσχόμενα μέτρα και παράλληλα θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι θα είναι πολύ δύσκολο και στο μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερβεί τους εσωτερικούς της διχασμούς περί Ρωσίας. Αυτό είναι μια διαδικασία που θα πάρει χρόνο. Νομίζω όμως ότι η εταιρική σχέση προς Ανατολάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση γιατί γεφυρώνει αν θέλετε τα χάσματα εντός της Ένωσης και παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στις ε, ανεπίλητες σειράξεις, θεωρώ ότι θα έχει θετικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των σειράξεων στην περιοχή αυτή. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία ακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής σας που με καλέσατε σήμερα για να σας μιλήσω σχετικά με τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νότιο Καυκάσου. Προτίθεμαι να σας κάνω μια ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Καύκασο το 2009 και να σας πω πού ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την παρουσίαση λοιπόν θα ήθελα να εστιάσω στην περιφερειακή επέμβαση και τι συμβαίνει σε περιφερειακό επίπεδο στον Νότιο Κάφκασο. Και επίσης θα σας πω πού βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιες σκέψεις σχετικά με το τι προσθέμενη αξία μπορεί να προσθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την οικοδόμηση της ειρήνης. Θα φροντίσω λοιπόν να είμαι σύντομη στην παρουσίασή μου από εδώ και δύο χρόνια όταν το Κοινοβούλιο ε, ψήφισε το έκθεση για το κάποιο το 2008 η κατάσταση έχει αλλάξει ιδιαίτερα μιλήσω για την κατάσταση που επικράτησε μετά τον Αύγουστο 2008 γνωρίζετε την κατάσταση πολύ καλά αλλά ήταν με ένα σημείο καμπής και οδήγησε σε μεγάλη... Μια κατάσταση πολύ πιο ασταθή και λίγο πολύ ξεπάγωσε όπως λέμε συχνά στην ορολογία της Στοκχόλμη στην ε, σύρεξη στην περιοχή. Όμως το 2008 δεν ήταν το μόνο αρνητικό. Στο 2008 δεν είχαμε τις μόνες αρνητικές εξελίξεις και από τότε και το 2009 δεν βελτιώθηκε πολύ η κατάσταση. Η Ρωσία παραμένει σε καθεστώς παραβάσεως των ε, συμφωνιών κατά παυστού πυρός του Οκτωβρίου του 2008. Δηλαδή δεν έχει αποσύρει σε επαρκή αριθμό και δεν έχει ε, φέρει στα μετόπιστα τα στρατεύματά της. Δεν τα έχει μετακινήσει. 5.000 στην Νότια Οσετία και άλλους 5 στην Απχαζία έχει ακόμα. Έχει μάλλον αυξήσει τις, ε, τα στρατεύματά της στις μη αναγνωρισμένες ε, περιοχές, μη αναγνωρισμένους θύλακες. Έτσι λοιπόν ε, εντάσσονται ε, δεν εντάσσονται πλέον σε διεθνείς δυνάμεις, δεν είναι διεθνείς στρατεύματα της ε, ΚΑΚ ή άλλης οργάνωσης, αλλά μόνο ρωσικά στρατεύματα. Και έτσι αλλάζει βέβαια σημαντικά η κατάσταση στην περιοχή. Επιπλέον η Ρωσία φαίνεται πώς προγραμματίζει τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις στην Απχασία και την Νότια Οσετία, εννέα, ε, εννέα ετή προγράμματα, 500 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση των ε, συνόρων και της παρουσίας τους εκεί και φαίνεται ότι σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατιωτική βάση στην Απχασία και μάλιστα στην Ουμτσανσίρα της ε, Μαύρης Θάλασσας, ίσως ήδη να σκοπεύουν να εγκαταστήσουν τέτοια βάση που να αντικαταστήσει αυτή τη Σεβαστουπόλου. Τουλάχιστον αυτό είναι οι αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι μάλλον απίθανο. Γιατί δεν έχει αρκετά βαθιά ύδατα η Νούμσανσίδα ε, σε σχέση με την Σεβαστούπολη ώστε να αποτελέσει ένα αρκετά μεγάλο λιμένα και βάση ναυτική, αλλά πάντως ε, οι φήμες εκεί πηγαίνουν. Αυτά. Ω προς την ε, προετοιμασία τη Ρωσία για τι μακροπρόθεσμες εξελίξει. Επίση, είδαμε ότι έκλεισε η ΟΑΣΕ την αποστολή τη, τα Ηνωμένα Έθνη, την αποστολή προ το 2009. Μας έγινε μόνο το UMMM που ε, διαδραματίζει ε, σημαντικό ρόλο βέβαια στη γεωργία, αλλά δεν έχει πρόσβαση ή πολύ περιορισμένη θα έλεγα πρόσβαση στην Απχαζία και την Νότια Οσετία. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ τώρα, άλλη περιοχή σύγκρουσης ε, στο Νότιο Κάφκασο, δεν παρουσιάζει εξελίξεις. Η κατάσταση ω προς την ασφάλεια επιδεινώνεται. Το 2009 συνεχίζονται οι παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, χρησιμοποιούνται πιο βαριά όπλα, ε, οβίδες, ε, ελεύθεροι σκοπευτές επίσης χρησιμοποιούνται, όλοι μη χρησιμοποιούνται. Πολύ λίγες εξελίξεις έχουμε ή τουλάχιστον λίγες θετικές εξελίξεις. Με αυτή λοιπόν την ε, μάλλον αρνητική εικόνα ε, θα έλεγα ότι σε περιφερειακό επίπεδο λίγες είναι οι θετικές εξελίξεις. Το μόνο που θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ως μια ακτίδα φωτός στην περιοχή ευρύτερα είναι η υπογραφή των πρωτοκόλων μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας τον Οκτώβριο του 2009. Η υπογραφή των πρωτοκόλων αυτών δεν συνέβη από τη μια μέρα στην άλλη, όπως καταλαβαίνετε. Ε, δεν ήταν κεραυνός ενεθρία, ήταν αποτέλεσμα πραγματεύσεων πολυετών που διευκόλυνε η Ελβετία και που έφεραν έτσι την Τουρκία με την Αρμενία στο σημείο τη υπογραφής των πρωτοκόλων, αλλά ταυτόχρονα σηματοδοτείται και μία δεκαετία ε, προσέγγισης μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών και απλών ανθρώπων. Είναι κομμάτι μιας διαδικασίας λοιπόν, ε, διαδικασίας επεδοκοινωνιών των δύο κρατών που μας έφερε σε ε, στο σημείο της υπογραφής των πρωτοκόλων αυτών τον Οκτώβριο του 2009. Τρία εις βασικούς σκοπούς εξυπηρετούν τα πρωτόκολλα αυτά, αναπτύσσουν διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας, ανοίγουν ε, τα σύνορα που είναι κλειστά εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα μεταξύ των δύο χωρών και θεσπίσουν διμερείς ε, επιτροπές, η μία μάλιστα θα ασχοληθεί με την ιστορική διάσταση, τα, τα ιστορικά προβλήματα μεταξύ των δύο κρατών αυτών. Φυσικά όλα αυτά θα είχαν συμβεί χωρί τη ρητή στήριξη της ε, Ρωσίας. Πράγμα το οποίο να εκπλήξει κάποιους ε, που γνωρίζουν την ε, ιστορία της Ρωσίας και της τάστης την παραδοσιακή. Η, Ρωσία όμως διευκόλυνε αυτή την προσέγγιση και για λόγους οικονομικού συμφέροντος, γιατί θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει ε, το άνοιγμα των συνόρων, θα μπορούσε να διευκολύνει τις επενδύσεις της Ρωσίας στην Αρμενία, θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι δυνατότητες για πρόσβαση της Ρωσίας στην αρμενική βάση ε, πρόσβαση και μεταφορά εξοπλισμού, δυνατότητες εμπορικών συναλλαγών με την Τουρκία και την Λιβύη περιφέρεια. Και ενδιαφέρον είναι ότι η Ρωσία υποστήριξε αυτή την κίνηση, αυτή την προσέγγιση. Είδαμε δε ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια μια σαφέστατη εντατικοποίηση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας Βέβαια, μεγάλο τμήμα τη οικονομία και των σχετικών συναλλαγών συνδέονται με τον τουρισμό και πέρυσι οι τουρίστε από τη Ρωσία ήταν η μεγαλύτερη ομάδα τουριστών που επισκέφθηκε τη Ρωσία. Επίση, υπάρχουν σαφέστατα κοινά συμφέροντα. Πρόκειται δηλαδή για συμφωνίε για, το, για το South Stream, το νότιο ρεύμα ή την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα για τον αγωγό South Stream ε, ή άλλα τέτοια ζητήματα. Η πρόσβαση δηλαδή, που προσφέρει η Τουρκία στη Ρωσία για τους αγωγούς ή η συμφωνία για την ανάπτυξη ενός κοινού ομίλου, ε, ε, μια σύμπραξη κοινή για, ε, για τον αγωγό του, της Αμψούντας Τζιχάν και άλλα τέτοια ενεργειακά σχέδια που όμως δεν είναι τα μόνα που φέρνουν πιο κοντά την Τουρκία με τη Ρωσία. Πριν από δύο εβδομάδες ακόμη ήταν ο Πρωθυπουργός Ερντοάν σε επίσκεψη στη Ρωσία. Ε, προσέφερε τη δυνατότητα της κατάρρισης των απαιτήσεων για θεώρηση διαβατηρίου στη Ρωσία και μάλιστα πρότεινε να αρχίσουν οι δύο χώρες να, κάνουν κοινέ υπουργικέ συναντήσεις. Να συνεδριάζουν από κοινού τα υπουργικά συμβούλια. Πράγματα λοιπόν τα οποία δείχνουν ότι οι δύο αυτές χώρες ήταν χωρισμένες από το ε, σιδηρούν παραπέτασμα και τον ψυχρό πόλεμο όλα αυτά τα χρόνια, τώρα αρχίσουν και ε, συσπυρώνονται και ενώνουν τι δυνάμει του Νότιου Νότιο Κάφκασο. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε ω απειλή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει μάλλον να εξετάσει τι δυνατότητε, να αξιοποιήσει τι δυνατότητε που προσφέρονται στην περιοχή, τι νέε δυνατότητε, τι νέε ευκαιρίε και νέε δυνατότητε για συνεργασία, για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Ε, προφανώς θα προχωρήσει μακροπρόθεσμα αυτή η νέα συμμαχία μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Είναι τέτοια η επένδυση δυνάμεων και κόπων που δεν μπορεί να είναι πρόθεσμα αυτή η προσπάθεια. Αυτό που είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες ιδιαίτερως είναι ότι η προσέγγιση Τουρκίας-Αρμενίας δεν πάει καλά. Ε, βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει και κολυσιεργία και εκεί που περιμέναμε ότι θα υποβληθούν για έγκριση στα ε, εθνικά κοινοβούλια της Τουρκίας και της Αρμενίας αντίστοιχα τα δύο πρωτόκολλα και ότι θα εκφραστεί υποστήριξη ε, για την κύρωσή τους, φαίνεται μάλλον ε, ασθενικό το ενδεχόμενο αυτό. Ε, ανάβουν τα αίματα στις ε, δηλώσεις και τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας και φαίνεται ότι η Τουρκία αρχίζει να ξανασκέφτεται τη στάση της και οι ρεάλ πολιτικοί και οι παραδοσιακές αντιδράσεις έχουν πάρει το πάνω χέρι. Υπάρχουν μερικές φορές και ισχυρισμοί πως η Τουρκία ε, πρέπει να υποστηρίζει τους αζέρους αδελφούς της για λόγους ιστορικούς, εθνικούς ε, και ε, θρησκευτικούς, αλλά εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο επανέρχεται ως προς τις συμφωνίες με την Αρμενία, αλλά μάλλον οικονομικοί οι λόγοι. Τον Οκτώβριο όταν υπέγραψε τα πρωτόκολλα η Ρωσία με την Αρμενία ήταν κατά τύχη η ίδια μέρα κατά την οποία το Αζερβαϊτζάν υπέγραφε ε, σύμβαση με την Ρωσία για μεταφορά φυσικού αερίου. Ήταν δηλαδή η εποχή όπου η Τουρκία ανησυχούσε για το κατά πόσον θα ε, έχει προβλήματα ως προς τη μεταφορά ε, αερίου από το οποίο εξαρτάται τόσο πολύ και από το που θα περούν οι αγωγοί του αερίου. Αισθανόταν την ανησυχία ότι δεν θα εξασφαλίσει τόσο εύκολα το φθηνό αζέρικο φυσικό αέριο. 120 δολάρια τα χίλια κυβικά μέτρα κοστίζει αυτή τη στιγμή για την Τουρκία το φυσικό αέριο του Αζερβαϊτζάν. Έτσι λοιπόν το ζήτημα της προσέγγισης Αρμενίας και Τουρκίας έχει φτάσει σε ένα σημείο στασιμότητας με αρνητικές ε, επιπτώσεις φυσικά, ενδεχομένως και ως προς την επίλυση της σύγκρουσης των Κορνοκαταπάχ Καταπάχ. Τα δύο αυτά ζητήματα είναι αλληλένδετα, δεν μπορούμε να το λησμονούμε και αλληλοεξαρτώμενα. Ταυτόχρονα όμως μπορούν να προχωρήσουν και εκ παραλίλου. Έτσι λοιπόν, εάν ε, βραδιπορήσει η προσέγγιση μεταξύ Τουρκία και Ερμενία, κατά πάσα πιθανότητα και η διαπραγματεύση για τον Ακόρνο Καραμπάχ θα ε, καθυστερήσουν ή θα σταματήσουν. Για, τις για ΗΠΑ θέλω να σημειώσω ότι μειώνεται σταδιακά, παρατηρείται μια σταδιακή μείωση της παρουσίας των Αμερικανών στην περιφέρεια και για την ε, Γεωργία, όπου είχαν διαδραματίσει η επικυβέρνηση Σμπούχ πολύ ενεργό ρόλο, αλλά και για την επίλυση της διαφοράς των Αγκόρνο Γαραμπάχ. Ε, τώρα τι θέση μένει ε, τι ρόλο μένει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προκειμένη κατάσταση. Μπορούμε να έχουμε τρεις διαφορετικά, τρία διαφορετικά πεδία δράση. Καταρχά, πολύ πιο σαφή περιφερειακό ρόλο. Με την εκκίνηση τη Ανατολική Εταιρική Σχέση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε ένα πολύ σημαντικό βήμα και χειρονομία ε, συμμετοχή στην περιφερειακή πολιτική και ιδιαίτερα τις περιφερειακές πλατφόρμες που θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία τους για την επίλυση των περιφαριακών ε, διαφορών και σειράξεων. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσει να παίζει τον ε, ρόλο του η μάντα μεταφορά η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την επικοινωνία μεταξύ αυτών των περιφερειακών ε, χώρων ή πλατφορμών. Πρέπει να, υπο... να μην περιμένει δηλαδή τις εξελίξεις από μόνες τους να προχωρήσουν, αλλά να τις στηρίξει και να υποβοηθά τις πλατφόρμες στην προσπάθειά τους για επικοινωνία και επίλυση των διαφορών. Επίσης, ήθελα να σημειώσω ότι μπορεί η Συμφωνία τη Λισαβόνα. Ε, η συνθήκη πρέπει να είναι η ομιλήτρια, ε, προσφέρει νέα μέσα και δυνατότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα θεσμικά της όργανα, πάλι χρειάζεται κάποιο συγκεκριμένο, κάποια συγκεκριμένη παρουσία ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιο συγκεκριμένο εκπρόσωπο δηλαδή που θα διαδραματίσει όπως ήδη συμβαίνει ένα ρόλο εκπροσώπου και μετά τη θέση ισχύ της Συνθήκης Λισαβόνας. Επίσης στην ομάδα της OMC όταν αποχωρήσει ο ε, πρεσβευτής ε, Φασιέ ίσως θα πρέπει να υπο... Ε, ίσως θα πρέπει να αναθεωρηθεί ο έντονος ρόλος που παίζει η Γαλλία στην περιοχή αυτή. Και βεβαίως θα πρέπει να εξετάσουμε με ποιο τρόπο θα υποστηρίξουμε την υπόθεση του Νακόρνο Καραμπάχ, είτε μέσα από την αποστολή της ΟΑΣΕ που έχουμε μόνο έξι παρατηρητές, ή με νέα παρουσία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. Πάντως πρέπει να συνεχίσουμε να προσφέρουμε οικονομικέ προοπτικές για τις ε, περιοχές για τις χώρες περιοχής, έχουμε ε, γενικές συμφωνίες, ε, μεγάλες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο για συμφωνίες σύνδεσης και νομίζω ότι για να μπορέσει πραγματικά να διδραματίσει το ρόλο που πρέπει να τέτοια συμφωνία, δεν θα πρέπει να αποκλείει το ενδεχόμενο της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του δένα τρόπο. Φαντάζομαι βέβαια ότι είναι δύσκολο να υποστηριχθεί κανείς ρητά ε, την δυνατότητα της προσχώρησης από τα κράτη αυτά, αλλά δεν θα πρέπει και να την αποκλείσει. Ούτε, να την υποσχεθούμε, ούτε να την αποκλείσουμε δηλαδή. Επιπλέον, πέραν του, διμερ, του πολυμερούς έχει και διμερές, ε, διμερείς σχέσεις και διμερεί ρόλο να διδραματίσει με αυτές τις μη αναγνωρισμένες οντότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα με την ε, Νότια Οσετία και την Απχαζία και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της ε, με την παρουσία της, έντονη παρουσία και ανάμειξη στις, ε, στην περιοχή με τις μη αναγνωρισμένους θύλακες, ε, ίσως και με το Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία θα ήταν σκόπιμο να συνεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν της ε, Νότιας και της Αφχαζίας δηλαδή, για να δει πώς θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος του Νακόρο Καραμπάχ. Επίσης θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ε, ως βασική αρχή ε, τηρούμε την, την αναγνώριση της εδαφικής ακαιρεότητας όλων των κρατών του Νότιου Καυκάσου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε στις διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην Νότια Σετία, Απχασία και τον Ακόνο Καραμπάχ. Εν τέλει, άλλο σημαντικό στοιχείο που θα μπορούσε να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν να ξεκινήσει ε, διαπραγματεύσει σε πολλαπλά επίπεδα, δηλαδή όπως έκανε άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνέχιση των ε, συνομιλιών της Γενέβης, ε, όπως και και μέσα από τη μορφή των συνομιλιών του Ναγκόρνο Καραμπάχ, ταυτόχρονα όμως αναλογιζόμενοι και το πώς θα μπορούσε να τι είδου συνέχεια θα μπορούσε να δοθεί στι συνομιλίε. Στι συνομιλίε δηλαδή θα πρέπει και να επιτρέπουν την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών, αλλά δεν θα πρέπει να σημάνουν επικοινωνία μόνο με του Αζέρου και του Αρμένιου, αλλά και με ε, του Αζέρου του Ναγκόρνο Καραμπάχ και με του Αρμένιου του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αυτά είχα να πω μέχρι τώρα. Ίσως θα ήταν καλό να λάβει το λόγο τώρα ο συνάδελφος κύριος Κόεν. Η κοινωνία των πολιτών όμως, κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι έχει διαδραματίσει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στο παρελθόν και τώρα στο παρόν και στην Νότιο Σετία και στο, στην Απχασία και στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Μας ενδιαφέρει ο διάλογος με την ε, κοινωνία των πολιτών για την ανοικοδόμηση της ειρήνης. Φυσικά δεν μπορεί να κάνει τα πάντα η κοινωνία των πολιτών. Δεν μπορεί να, δηλαδή να προσφέρει ή να φέρει την ειρήνη σε μια περιοχή, αλλά μπορεί να είναι παρούσα την ώρα που συνάπτεται η συμφωνία ή άπαξ και συναυθεί η συμφωνία, ώστε να θέσει σε κίνηση, σε λειτουργία όλη τη διαδικασία. Το τα πράγματα όμως πάνε στραβά, όπως είδαμε πρόσφατα με την Τουρκία και την Αρμονία, μπορεί, μπορεί και πάλι να βοηθήσει σε περίπτωση που αποτυγχάνουν οι διαπραγματεύσεις για την αποκατάσταση κατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας. Ε, και σε αυτό το ρόλο μπορεί πολλά να προσφέρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δόκτωρ Κόεν έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να σας μιλήσω σήμερα. Δύο πράγματα θέλω να αναφέρω ξεκινώντα. Καταρχάς να σας πω κάποιες ιδέες ως προς τη φύση και τα κοινά χαρακτηριστικά των συγκρούσεων και δεύτερον, αναφερθώ στα προβλήματα και τις ευκαιρίες ως προς τη δυνατότητα να τη των, της περιφέρειας, τις ε, κοινωνίες και το ρόλο βέβαια ή τα διδάγματα μπορούμε να αποκομίσουμε από το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε ό,τι συμβαίνει στην περιοχή, ούτως άλλως είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση, αλλά βεβαίω αν έχετε συγκεκριμένε ερωτήσεις, πολύ ευχαριστώ να δώσουμε τις απαντήσεις που μπορούμε. Ως προς το, τα ευρύτερα ζητήματα που μπορούμε να εντοπίσουμε ως αίτια της σύγκρουσης. Θα ήθελα να σημειώσω ότι όταν μιλούμε για συγκρούσεις στο Νότιο Κάφκασο, απαραίτητο είναι να ξεχωρίσουμε ότι πρόκειται για διαφορετικές συγκρούσεις. Δεν είναι τα χαρακτηριστικά του κοινά και δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κοινέ λύσεις και στις ε, τρεις αυτές συγκρούσεις, στις διάφορες συγκρούσεις είναι διαφορετικά τα δεδομένα, έστω και αν υπάρχουν περιφερειακοί σύνδεσμοι, συνδετική Κρήτη. Και όπως είπε στην άνθρωση Λορουρίτερα, δεν θα πρέπει να τις ονομάζουμε παγωμένες συγκρούσεις. Ήταν ε, λάθος επιλογή ο όρος αυτός και στο παρελθόν. Δεν ήταν ποτέ παγωμένες αυτές οι συγκρούσεις. Υπήρχαν δυναμικές εντάσεις στην περιοχή. Όμως αυτό που συνέβη με την... Ε, ε, και ξεπάγωσαν αυτές οι συγκρούσεις κατά κάποιο τρόπο είναι ότι έχασε η ειρηνευτική διαδικασία και οι διαπραγματεύσεις την νομιμοποίησή της στην περίπτωση όμως της Γεωργίας περισσότερο είδαμε ότι η Γεωργία έχασε την εμπιστοσύνη της στην ειρηνευτική διαδικασία, δηλαδή αποφάσισε ότι δεν μπορεί να της προσφέρει αποτελέσματα και έτσι αποφάσισε να ταράξει τα νερά, να αναλάβει μόνη της δράση, να φέρει το θέμα στο διεθνές επίπεδο και βέβαια με επικίνδυνα αποτελέσματα, με επικίνδυνες κινήσεις, γιατί μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρά τα αποτελέσματα, σε ένα βαθμό συνέβαλε στα όσα συνέβησαν τον, Αύγουστο του 2008. Και επίσης θα ήθελα να περάσω σε ένα άλλο πολύ σημασία ζήτημα που θα πρέπει να έχουμε τη Ρωσία. Η Ρωσία διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο και προκάλεσε και διατήρησε τις συγκρούσεις στην ε, ε, άμεση μετασοβιετική εποχή και στην ε, μη τήρηση το, της του πυρός το 1993 και ως τρίτο μέρος προσπαθώντας τόσο να μεσολαβήσει όσο και να στηρίξει κάποιο από τα μέρη των συγκρούσεων. Πάντως, εάν δούμε τη Ρωσία μόνο όσο τον ε, κατηγορούμενο στην υπόθεση αυτή, δεν θα καταλήξουμε πουθενά, γιατί θα πρέπει και τα συμφέροντα τη Ρωσία να κατανοήσουμε και να αναλάβουμε τι πρωτοβουλίε που θα μα επιτρέψουν να ε, συνεργαστούμε επικοδομητικά μαζί τη ε, και να μην την θέσουμε στο εδόλιο του κατηγορουμένου, γιατί αυτό θα μα βοηθήσει καθόλου στην επίλυση των διαφορών αυτών. Δυνατότητε και ευκαιρίε. Θα ήθελα να ξεκινήσω τώρα με την κοινωνία των πολιτών πρώτα απ' όλα, για τη δική μου προοπτική. Η είναι απαραίτητες τυπικές διαδικασίες ε, διαπραγματεύσεων, αν και όχι επαρκής, γιατί πάνω απ' όλα απαιτείται μια πιο ολιστική προσέγγιση για την εξέταση των διαφόρων πηγών και αιτιών ε, των συγκρούσεων και την εμπλοκή βεβαίως της κοινωνίας των πολιτών. Η αντίληψη που μπορεί να έχει το κοινό ή οι προσδοκίες ή και οι φόβοι σε σχέση με μια ειρνευτική διαδικασία παραμένουν αποκομμένες από την περιορισμένη αλληλεπίδραση των πλευρών που κάθονται γύρω από ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Και όσο δεν έχουν επιληθεί αυτά τα ζητήματα, όσο δεν μπορούμε δηλαδή να επανευθαρμίσουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές με τις ε, ιδέες, τις συνείδηση, τις προσδοκίες των ε, πολιτών, δεν θα έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Και γι' αυτό εδώ είναι πολύ σημαντική συμπληρωματική ε, παρουσία της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και ο ρόλος της ως κινήτρου για πιο αποτελεσματική ε, πιο αποτελεσματικές προσπάθειες μέσα από τις διαπραγματεύσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν και να προσπαθήσουμε να εργαστούμε μαζί με την κοινωνία των πολιτών και να επιλύσουμε τις ε, ε, διαφορές. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα να γνωρίσουμε τον άλλον, να δώσουμε διαφορετικές εναλλακτικέ, να δώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις που θα διοχετευτούν στη συνέχεια στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και να βοηθήσουμε στις διάφορες προσπάθειες που θα οδηγήσουν σε, μετα... μεταστροφή στην αναλυτική συμπεριφορά και το πλαίσιο το ιδεολογικό που αποτελούν πολλές φορές την ίδια τη δομή μια σύγκρουση. Πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί με διάφορους τρόπους. Αν είχατε περισσότερο χρόνο, πολύ ευχαριστώ να σα δώσω και συγκεκριμένα παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η κοινωνία των πολιτών με τους φορείς που την εκπροσωπούν μέσα και έξω από την περιοχή να αναγνωριστεί ως ε, ουσιαστικός παράγων αλλαγής ε, και να σας παραδείγματα έχει μπορέσει να ε, ξεπεράσει τους φραγμούς και τους διχασμούς, έχει δημιουργήσει κοινά, ενδιαφέροντα και κοινό πεδίο συνομιλίας μέσα από τις τηλεοπτικές εκπομπές ή τις ε, πολιτιστικές εκδηλώσεις, έχει εξασφαλίσει ανάπτυξη αναλυτικής, επικοδομητικής ε, σκέψης μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και μέσα από διμερείς παρουσία παρουσίες έχει η κοινωνία των πολιτών δείξει πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από ότι τα κράτη που έχουν εμπλακεί σε αυτές τις ε, διαπραγματεύσει, και μάλιστα έχει μπορέσει η κοινωνία των πολιτών να κάνει τη δουλειά τη τόσο ήσυχα που δεν ε, φαινόταν καν στα μέσα μαζική ενημέρωση, και έτσι ήταν πολύ πιο αποτελεσματική. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ είναι τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, ε, που πολλές φορές όμως στην περιοχή τα βλέπουν με σφαλμένο πρίσμα και θα έλεγα όπως είχε πει ο Τζον Εφ Κένεντι παραφράζοντας τα λόγια του, μη σκέφτεσαι τι μπορείς να κάνεις για, το δικό σου, για τη δική σου πλευρά, για τη δική σου παράταξη, αλλά για την αντίπαλη παράταξη. Μόνο έτσι μπορείς να είσαι αποτελεσματικός. Αυτό σημαίνει μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη και αυτό νομίζω είναι πρέπει να επιδιώξουμε για την περιοχή. Επίσης πρέπει ιδιαίτερα να, δώσουμε, ε, να, να, να αναγνωρίσουμε ότι δεν μπορεί να ε, διχα, διαχωριστεί από την ε, καθημερινή πολιτική κοινωνία των πολιτών. Χρειάζεται η παρουσία της και η επίδραση της στην καθημερινή πολιτική. Και από τα όσα βλέπουμε σήμερα είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η μεταμόρφωση και επίλυση των διαφορών και συγκρούσεων ε, μέσα από την κοινωνία των πολιτών σημαίνει και μια συνενετική βάση και δομή υποστήριξης που δεν υπάρχει πάντοτε μέσα από τις παραδοσιακές δομές χρηματοδότησης ή παρέμβασης που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η διμερής χορηγή, γιατί μέσα από 18 μήνα επί παραδείγματι προγράμματα δεν μπορεί κανείς να φέρει την ειρήνη. Χρειάζεται πολύ ευρύτερο και πολύ πιο μακροχρόνιο πλαίσιο. Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και τα μέσα ή προσεγγίσεις που μπορεί να υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει πολύ μεγαλύτερη παρησία και να αναπτύξει την ε, ήπια δύναμη της ε, σε ευθυγραμμισμένη φυσικά με τι εξελίξει στον υπόλοιπο κόσμο για να βοηθήσει στην επίσημη των διαφορών. Όμω ε, η ήπια δύναμη δεν πρέπει να παραμείνει μόνο ε, στη θεωρία, γιατί δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Πρέπει να είναι πολύ πιο αποφασιστική και καθοριστική στα αποτελέσματά τη και ελπίζω να μπορώ να σα δώσω κάποιε συγκεκριμένε ιδέε. Υπάρχει παραδείγματι η ιδέα ότι ο εξευρωπαϊσμό είναι μια στρατηγική για την εξασφάλιση ε, επίλυση των διαφορών. Όμω αυτό αποτελεί μια εσφαλμένη αφετηρία. Ο εξευρωπαϊσμό δεν είναι απαραίτητα για ένα κράτο στόχο ή στόχος των οποίων μπορεί ε, ο πληθυσμός ενός αποσχιστέντος ε, μιας σα περιοχής εδαφών να προσυπογράφει και να επιδιώκει για να βοηθήσουμε αυτόν τον τρόπο στην επιλήτη αφορά. Αυτό ισχύει και για την Απχασία και για την Νότια Ζωτία και για τον Ακόρνο Καραμπάχ. Πέραν αυτών δηλαδή βλέπουμε ότι αυτές οι περιοχές και γιατί ε, είχαν ε, βρεθεί στο περιθώριο λόγω των δικών του στρατηγικών αλλά και των επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βρέθηκαν αποκομμένες και χωρίς διεξόδους και άρα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν οντότητε με διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Είδαμε ότι βλέπουν μάλλον αυτές οι περιοχές οι αποκομμένες, οι αποσχιστικές περιοχές, ότι αναγνωρίστηκε στο κοσφοπέδιο η ανεξαρτησία, αλλά παραδείγματι δεν δόθηκε δεν αναγνωρίστηκαν εξίσου οι δικές του προσδοκίε και αυτό βέβαια δημιουργεί προβλήματα εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρίσιμο λοιπόν στοιχείο θα είναι να επικεντρωθούμε στον τομέα του εκδημοκρατισμού και το τι μπορεί να προσφέρει ο εκδημοκρατισμός ε, στο στόχο μας. Ο εκδημοκρατισμός και η δημοκρατία είναι όρος αναγκαίος αλλά όχι επαρκής ε, για την αντιμετώπιση αυτών των ε, συγκρούσεων που γνωρίζει ο Κάφκασος η εξαγωγή δημοκρατικών εκλογών στις χώρες περιοχής, που έχουν όμως ε, προβληματικά δικαστικά συστήματα και ελλειπείς δημοκρατικές δομές, δεν μπορεί να αποτελεί επαρκή ε, στόχο. Η προαγωγή της δημοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης πρέπει βεβαίως να μειώνει τα κενά και τα χάσματα που τους, τις διχαστικές γραμμές μεταξύ των πληθυσμών των περιοχών αυτών και θα πρέπει βεβαίως να, δώσουν, να κάνουμε προσπάθειες προς το στόχο αυτό, αλλά η απομόνωση των 15 ετών δεν έχει μπορέσει να φέρει ε, λύσεις στις, ε, στα προβλήματα, ούτε έχει επιτρέψει τον επαναπατρισμό ε, των, ε, των εκτοπιστέντων. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να αναζητήσουμε άλλες στρατηγικές για να επιδιώξουμε τους στόχους μας. Στη Γεωργία, παραδείγματι, τώρα αναπτύσσεται μια νέα σημαντική στρατηγική για την προαγωγή της επικοινωνίας με την Απχασία και την Νότια Οσετία. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να αναφερθεί και σαν στόχος η αποχώρηση των στρατευμάτων ε, η αποχώρηση μάλλον των κατεχόντων τα εδάφια αυτά, πράγμα το οποίο δεν είναι απαραίτητο μπορούμε, δεν είναι δεδομένο ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε και εμείς και ταυτόχρονα δεν μπορούμε να, ε, δεν, δεν είναι σωστό να απευθύνουμε κατηγορίες συνέχεια στη μία πλευρά ε, στα αποσχιστέντα εδάφη δηλαδή, ε, σαν να είναι αυτά υπεύθυνα για τα πάντα. Με την Απχασία ιδιαίτερως βλέπουμε ότι πρόκειται για μια συνεχιζόμενη και ενεξελίξη πολιτική διαδικασία και ταυτόχρονα είτε μας αρέσει είτε όχι, οι αρχές της χώρας όταν τις απομονώνουμε είναι λιγότερο δεκτικές οποιαδήποτε υπόδειξη και επίσης η κοινωνία των πολιτών στις περιοχές αυτές παραμένουν ε, εκτεθειμένες και κλειστέ στα δικά μα μηνύματα γιατί βλέπουν ότι μόνο τι κατηγορούμε και δεν έχουν καμιά ελπίδα για επικοινωνία με τον έξω κόσμο το οποίο δεν διευκολύνει καθόλου την, ε, τις προσπάθειες για την ειρήνη και την ασφάλεια. Ίσως θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ πιο θαραλέοι αλλά και φάνταστοι στην προσέγγισή μας. Ε, ακούσαμε να γίνεται λόγος για, πολύ, για το πολύ σημαντικό σύνθημα ε, εμπλοκή αλλά όχι αναγνώριση, engagement but not recognition και πρέπει να αναλογιστούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Οι πολιτικοί ηγέτες και κατά προτίμηση δημοκρατικά εκλεγθέντες ε, εκπρόσωποι των λαών τους θα πρέπει βέβαια να επιδιώκουν ειρηνικές ε, ε, λύσεις στα προβλήματα, αλλά δεν έχουν προωθήσει ιδιαίτερα στις ηγέτες των περιοχών αυτών τις λύσεις που θα μπορούσαν να συνεπάγονται και την αποδοχή συμβαστικών λύσεων και να οδηγήσουν στη συνέχεια στην επίλυση των διαφορών, ίσως γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν το εσωτερικό τους έρισμα και την εσωτερική τους ισχύ. Ίσως εδώ μπορεί η κοινωνία των πολιτών να διαδραματίσει το σημαντικότερο ρόλο ενδεχομένω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εν προκειμένου θα μπορούσε να διαδραματίσει τον εξή ρόλο και να δείξουμε, όπως είπα νωρίτερα, την εμπλοκή μας και να δώσουμε εφάνταστες λύσεις, αλλά και ταυτόχρονα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν πολύ σημαντικούς πολιτικούς ε, περιορισμούς ή περιορισμούς ως προς την αντίληψη των καταστάσεων και των λύσεων. Δηλαδή δεν έχουν επαφή με τα αποσχιστέντα απομονωθέντα αυτά εδάφη, ε, δεν μπορούν ε, να, ε, να αγνοήσουν τα προβλήματα και τις σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων στην προσπάθεια για επαφή και συνεργασία με τις κυβερνήσεις οι οποίες βρίσκονται στην εξουσία. Ε, και μερικές φορές είναι υπερβολικά επιφυλακτικές οι αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις ε, κινήσεις και, τις, ε, και τη στάση τους. Ίσως θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι έχουν αρκετά μεγάλη ευθύνη ως προς την επίλυση των διαφορών και πολύ μεγαλύτερη από ότι οι, Ηνωμένε Πολιτείε, η ΟΑΣΕ ή η Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φροντίσει να μην πέσει στην ίδια παγίδα που έπεσαν οι άλλοι διεθνείς παράγοντες που έμπνεπλάξαν στις φορές αυτές. Ε, πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να γνωρίσουμε ότι είναι πολύ ε, λεπτή η κατάσταση, ευάλωτη, ε, εύθραυστη καλύτερα και επίσης ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε στην κοινωνία των πολιτών να αναλάβει το ρόλο της, να σπάσει τα ταμπού και να ανοίξει ορίζοντες ε, έτσι ώστε να βοηθήσει την αλλαγή των δεδομένων μιας σύγκρουσης. Η γεφύρωση των χασμάτων, ίσως να μην μπορέσει να δώσει τα αποτελέσματα που θα ήθελαν ειδικά η Γεωργία και το Αζερπαϊτζάν αλλά ίσως να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ε, διαφορών. Δεν είναι μονολυθική η προσέγγιση και δεν μπορεί να είναι μονολυθική. Χρειάζεται μια αλλαγή μέσα από τις κοινωνίες οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί θα πρέπει να ε, ενθαρρύνουν ε, την κοινωνία των πολιτών να δραματίσει το ρόλο της και όχι να προσπαθούν να την ελέγξουν και η κοινωνία θα πρέπει από πλευρά της να μάθει ότι έχει καθήκον και να ελέγχει τις κυβερνήσεις της αλλά και να συνεργάζεται μαζί τους και ένα τελικό σχόλιο η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη εν γένεια πιστεύω έχει να κάνει μια επιλογή ως προς την αντίληψη της για τα πράγματα δηλαδή αν η ειρήνη είναι όρος για την αλλαγή ή αν η ειρήνη είναι όρος για τη σταθερότητα. Και το πρόβλημα που είχαμε πάντοτε στην περιοχή αυτή είναι ότι ανταποκρινόμαστε μόνο σε κρίσεις, δηλαδή προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε σταθερότητα και όχι να μετατρέψουμε τις ε, συγκρούσεις σε όρο της ειρήνης και πέραν αυτής της μακροχρόνιας ειρήνης. Ευχαριστώ. Grazie. Quindi procediamo a questo punto a raccogliere le domande che verranno dai colleghi. Θα ακούσουμε τώρα τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Θα τις ομαδοποιήσουμε δύο-δύο για να μπορούν να απαντήσουν και οι καλεσμένοι μας. Πέτερλε και Σέβερινγκ έχουν στήσει το λόγο. Πέτερλε. Ευχαριστώ και τους τρεις ε, ομιλητές ε, για τις ε, τόσο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Θα ήθελα να πω ότι έχω μια προκλητική ερώτηση. Μόνο ότι πολλές από τις προτάσεις που έγιναν σχετικά με την επίλυση αυτών των σειράξεων έχουν ήδη διαγραφεί. Θα ήθελα να πείσω την κυρία ποια θα ήταν τα πρώτα βήματα σε περίπτωση που θα αναλάβανε αυτή το ρόλο της Λέδης Άστον. Ε, ε, Σέβεριν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Μερικές ερωτήσεις έχω. Πρώτον, πιστεύετε ότι αυτές οι σειράξεις αποτελούν ένα κομμάτι, αποτελούν διάφορα κομμάτια μιας συνολικής κρίσης στη σχέση τους με την Ρωσία στη νέα διεθνή τάξη και εφόσον δεν διευκρινιστεί αυτό το καθεστώς τότε θα είναι πολύ δύσκολο για την Ρωσία να μπορέσει να συμμετάσχει στην επίλυση αυτών των κρίσεων. Σημείο 2. Επανειλημμένα και όχι μόνο εδώ στον οίκο μας, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΣΑ, συζήτησαν γιατί με την αναγκαιότητα ή την δυνατότητα να προσφέρουν στο Νότιο Κάφκασο ένα σύμφωνο σταθερότητας το οποίο θα ρυθμίζει και τα ζητήματα των ε, παγωμένων αυτών σειράξεων και τη δυνατότητα ε, ένταξης των αποσχιστέντων περιοχών. Τι πιστεύετε λοιπόν σχετικά με αυτήν την πιθανότητα και κάτι ακόμα, έχουμε συζητήσει και σε διάφορες εκθέσεις του Κοινοβουλίου έχουμε συμπεριλάβει την ιδέα της ανάγκης μιας διάσκεψης για την ασφάλεια και τη συνεργασία στον Νότιο Κάυκασο. που θα εξετάσει παράλληλα και το ζήτημα της ε, ουδετερότητας ε, της περιοχής προκειμένου να επιλθούν κάποιες ε, διαμάχες που υπάρχουν στην περιοχή. Και τέλος είπατε ότι πρέπει να αφήσουμε ανοιχτέ τις θύρες για τη δυνατότητα πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτών των χωρών. Ειλικρινά πιστεύω ότι αυτό ε, δεν είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση. Πολύ αμφιβάλλω γι' αυτό. Δεν θα ήταν πιο ρεαλιστικό να μην τους προσφέρουμε μεν ένταξη, αλλά ε, το ευρωπαϊκό μοντέλο έτσι ώστε να μπορέσουν να εγκαθιδρύσουν σε εκείνη την περιοχή ένα είδος κοινοπολιτείας ε, ένωσης ε, των κρατών του Νοτιού Κάφκασου. Ευχαριστώ. Οι εισηγητές. Παρακαλώ. Ποιος θα ξεκινήσει. Πολύ σύντομα να πω κάτι θα αφήσω τα υπόλοιπα στους συναδέλφους, αλλά θα έλεγα πως ε, πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη υπόμονη. Είναι ένα θέμα ιδιαίτερα περίπλοκο και δεν μπορούμε να κάνουμε άμεσα αλλαγές. Τώρα για τις ε, παγωμένες ε, σειράξεις Παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον όρο frozen conflict γιατί δεν μας βοηθάει. Τώρα, εάν αποτελούν κομμάτι μιας ε, γενικότερης κρίσης, ναι, νομίζω ότι η Ρωσία παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το ζήτημα, αλλά θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το πλαίσιο. Αυτό που προκαλεί τις σειράξεις έχει άμεση σχέση pre-Soviet trend, and it linked to issues that would be part το γεγονό είναι πώς, τι σχέση επιθυμεί να έχει η Ρωσία με, τις, ε, με τα κράτη αυτά. Εδώ υπάρχουν διάφορες προκλήσεις σχετικά με την ταυτότητα, την πρόσβαση σε ε, πόρους. Ε, υπάρχουν διαφορέ σε ό,τι την αντίληψη με το, για το παρελθόν. Σε μια περιοχή σαν αυτήν υπάρχουν και προβλήματα με την ε, με τις μειονότητες, την αυτοδιάθεσή τους κλπ. απέναντι στα πρώην Σοβιετικά κράτη. Σίγουρα υπάρχει κάποια ιεράρχηση ανάμεσα σε αυτά τα προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να ξεφύγουμε από μια τέτοια νοοτροπία για να μην θεωρούμε ότι η Ρωσία αποτελεί το πρόβλημα Η Ρωσία είναι σαν τον ήλιο στην έρημο, θα συνεχίσει να λάμπει. Πρέπει λοιπόν να τα βρούμε και να... για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Έχουμε το, μιλάμε για τον Νότιο Κάφκασο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Βόρειο Κάφκασο είναι μια περιοχή που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Νότιο Κάφκασο. Τώρα η Απχαζία έχει αλλάξει την κατεύθυνσή της σε ό,τι φορά με την Γεωργία. Και προβλήματα στον Βόρειο Κάφκασο σίγουρα θα έχουν αντίκτυπο στον Νότιο Κάφκασο. Λοιπόν, δημιουργώντας ε, μια αυθαίρετη κοινότητα με τις χώρες αυτές του Νότιου Κάφκασου δεν θα ήταν ορθό σε αυτή την περιοχή τα κράτη αγωνίζονται να ανακτήσουν την ταυτότητά τους και νομίζω ότι δεν είναι διατεθειμένοι να υπαναχωρήσουν το γεγονό ότι για να διανύσει κανείς 100, μίλια θα πρέπει να κάνει παρακάμψεις χιλίων και πλέον μιλέων ε, είναι πρόβλημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό έχει επίπτωση στο εμπόριο, στην ε, διακίνηση. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν αυτές οι, αυτές οι δομές. Υπάρχουν ελάχιστες πολιτικές δομές. Υπήρχε η πρωτοβουλία του Γρηγορίου του για να Νοτιού Καυκάσου, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί το να μην πιέσουμε τις εξέλιξεις. Το, το σύμφωνο για σταθερότητα του Νοτιού Κάφκασου είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω πως η περιοχή είναι έτοιμη να το δεχθεί σε αυτή τη φάση. Και τέλος, σε ένα σύντομο σχόλιο για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην περιοχή και την ε, στρατιωτική ουδετερότητα. Νομίζω πως ακόμα δεν είναι έτοιμη περιοχή. Αλλά το ζήτημα της, το, έχει μεγάλη σημασία διότι είδαμε ότι υπήρξε ένας ε, αγώνας ε, για τον εξοπλισμό. Είδαμε λοιπόν ότι σημαντικά κονδύλια επενδύθηκαν στην αγορά εξοπλισμού και όπλων και αυτό είχε, όπως καταλαβαίνετε, συνέπειες στην ευημερία του, των πολιτών. Αν μου ζητούσε η Λέδη Άστον τι θα πρέπει να κάνει, θα της πρότεινα τρία πράγματα. Καταρχάς, να στείλει τους συμβούλους της στην περιοχή και να μιλήσουν με όλους τους τοπικούς φορείς για να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και κατέστησε αφές από τις παρουσιάσεις του πάνελ γιατί είναι πολύ περίπλοκες διαφορετικές καταστάσεις που επικρατούν στις περιοχές αυτές. Κατά δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυρία Φρέιζερ το είπε στην παρουσίασή της, νομίζω ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και οι πολυμερείς πλατφόρμες, όλα τα μέσα, αυτά που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνουν στην Ένωση ευκαιρίες, τις οποίες θα πρέπει να αξιοποιήσει. Αυτό θα ανακύψει τα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να αξιοποιηθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο οι ευκαιρίες αυτές. Τρίτον, να εναρμονιστούν τα μέσα επιτόπου στην, στις Ένωσης υπό, στα πλαίσια της Συνθήκης Λισαβόνας. Αναφέρατε την στρατιωτική ουδετερότητα. Είναι δύσκολο το θέμα αυτό και ασφαλώς δεν είμαστε σε θέση να πούμε σε κυρίαρχα κράτη τι θα πρέπει να κάνουν ως προς την πολιτική τους. Αλλά συγκρίνοντας την κατάσταση στην Πρετνέστηρία, στη Μολδαβία και στη Γεωργία, Φυσικά το γεγονός ότι η Μολδαβία δεν έχει φιλοδοξίες για το ΝΑΤΟ έχει απαλύνει την οξύτητα της σύγκρουσης και έχει δώσει δυνατότητα στην Ένωση να συμμετάσχει. Αυτό παίζει ρόλο, αλλά παράλληλα αποτελεί και ένα πολύ δύσκολο θέμα. Επίσης επειδή, όπως αναφέρθηκε, τα κράτη αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα σε ό,τι αφορά θέματα κυριαρχίας. Και νομίζω ότι τα θέματα τα στρατιωτικά βρίσκονται στον πυρήνα της κυριαρχίας του κράτους. Τέλος, το θέμα των κρατών αυτών της κοινότητας διαμόρφωση μια μιας σχέσης κοινοπολιτείας με τις χώρες αυτές. Δεν νομίζω ότι αυτό θα ενδιέφερε τι χώρες αυτές. Δεν νομίζω ότι θα πετύχαινε το σχέδιο αυτό και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό όταν θα προσεγγίσει η Ένωση τα κράτη αυτά. Ο συνάδελφος Βόμποντα, ευχαριστώ. Για να επανέλθουμε στο τελευταίο αυτό στοιχείο στην απάντηση του κυρίου Κοέν προς τον κύριο Σέβεριν. Δεν έχω πιστεί απόλυτα, γιατί το, το 45-46 πολλοί έλεγαν ότι «Α, είσαι τρελός, Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τον πόλεμο». Δεν θα πρέπει να το ξεχάσουμε λοιπόν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος. έγιναν συνομιλίες στο Βερολίνο, στις οποίες και συμμετείχα σχετικά με το θέμα αυτό. Αν ζητήσουμε από τις χώρες να επικεντρωθούν στην ευημερία των πολιτών τους και στην οικονομική ευμάρεια, να χρησιμοποιήσουν πιο πολλά κονδύλια για τις υποδομές και λιγότερες, ε, λιγότερα κονδύλια προς το στρατιωτικό σκέλος, και ίσως να τους ενισχύσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα περιφερειακό, για παράδειγμα, στον Εύξηνο. Ίσως έτσι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια ιδανική εικόνα για μια οικονομική συνεργασία. Ας μην το αποκαλέσουμε ένωση σε πρώτη φάση. Και έτσι να εστιάσουμε την προσοχή πιο πολύ στην ε, ευημερία των πολιτών. Κάποιοι ηγέτες δεν το επιθυμούν αυτό ίσως, αλλά Ίσως προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Μικρές ερωτήσεις να σας κάνω. Ενημερώθηκα ότι στην ε, Γεωργία ξεκινάει η στρατιωτική εκπαίδευση στα σχολεία για να προετοιμαστούν για μια σύγκρουση. Αλλά ξέρετε, αυτή η προετοιμασία μπορεί να προκαλεί και ενδεχομένως πιο πολλές πιθανότητες για σύγκρουση για την Αρμενία και την Τουρκία, κυρία Φρέιζερ. Ίσως είναι κάπως ευθύνη της Τουρκίας που δεν επικύρωσε την συμφωνία. Αλλά από ό,τι άκουσα η Αρμενία λέει ότι αν η Τουρκία δεν επικυρώσει την ε, ε συνθήκη μέχρι κάποια προθεσμία, η Αρμενία θα κάνει και αυτή πίσω και θα υπαναχωρήσει ως προς την συμφωνία αυτή. Και φυσικά έχουμε το δύσκολο θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ και είναι σαφές ότι η Τουρκία δεν θέλει να χάσει εδάφη. Αλλά μιλήσατε πιο πολύ για την πλευρά την τουρκική. Τι γίνεται από πλευρά Αρμενίας. Και τελευταίο ερώτημα. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία. Ξέρει η αποστολή τι γίνεται στην Απχαζία και στην Οσοτία. Κάποιοι λένε ότι δεν έχουμε πρόσβαση, δεν έχουμε ελικόπτερα. Ε, άρα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ακόμα και αν υπάρχουν στρατιωτικές εξελίξεις στις δύο αυτές περιοχές, εμείς δεν θα το γνωρίζαμε. Και αυτό φυσικά θα ήταν πολύ επιβλαβές για οποιαδήποτε νέα αποστολή. Αν δεν ξέρουμε τι γίνεται και αν δεν έχουμε τα εργαλεία για να παρακολουθήσουμε τι γίνεται στην περιοχή αυτή. La Preda, il Preda, IPP. Merci infiniment. Je suis... Preda Θα κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Θα ήθελα να μάθω κάτι σχετικά με ένα από τα σημεία που αναφέρθηκε στον τίτλο δηλαδή η κατάσταση στην υπηρετητρία. Εντάξει, Νότιο Κάφκασο τα καταλάβαμε όλα. Η Περνιστερία όμως ως τμήμα της Μορδαβίας βρίσκεται ακόμα πιο κοντά μας. Σε μένα από το Βουκουρέστι απέχει τρία τέταρτα. Θα ήθελα να πω δύο, δύο πράγματα. Το ένα αφορά τη σχέση μας με τη Ρωσία, διότι η σχέση με τη Ρωσία, η Ρωσία επαναλαμβάνω, βρίσκεται πολύ κοντά μας. Γείτονα είναι. Η Ρουμανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα σε τρία τέταρτα ε, φτάνετε σε ένα σημείο που συναντάτε Ρώσους στρατιώτες. Εγώ υπήρξα μέλος αυτής του σώματος για την, με τις για την παρακολούθηση των εκλογών στη Μολδαβία και σε ένα έδαφος το ε, μολδαβικό πέφτω απάνω σε Ρώσους στρατιώτες. Εντάξει, πρέπει να μας λένε ότι πρέπει να είμαστε ε, δημιουργική, φάνταστη κλπ. Όλα αυτά πώς θα τα έχουμε, θα πετύχουμε όταν πέφτουμε πάνω στους Ρώσους στρατιώτες. Λοιπόν, σε... αντίθετα από το Νότιο Κάυκοσο έχουμε δύο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δήλωσαν πριν από την είσοδό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση πως πολίτες Μολδαβοί είναι πολίτες Ρουμάνοι αλλά και Βούλγαροι. Έχουμε και εδώ Βούλγαρους συναδέλφους που μπορούν να μας δώσουν στοιχεία. Ξέρω πως ε, κάποια στιγμή υπήρχαν περισσότεροι Μολδαβοί που γίνονταν Βούλγαροι από ότι Ρουμάνοι, συνήθω σημαίνει το αντίθετο, αλλά δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δεν συναντάται στην ε, Νότιο Κάφκοσο. Λοιπόν, πώς θέλετε να υπάρχουν αυτές οι σχέσεις με τις παγωμένες ε, σειράξεις που εμπεστώς δημιουργούν νέα πολιτικά δεδομένα στη Μολδαβία και δημιουργούν και εντάσεις το κάτω-κάτω. Χθες ένας ε, ανώτατος πολιτικό, ένα ανώτατο πολιτικό στέλεχος στη Μολδαβία είπε ότι φοβάται πως το σενάριο της ε, Γεωργίας θα επαναληφθεί ε, στην Μολδαβία. Πρόκειται για μια περιοχή που είναι στις θύρες της Ευρώπης. Δεν μιλάμε για Νότιο Κάφκασο εδώ. Ευχαριστώ. Άλλη μια ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ρωτήσω τους ομιλητές για την, ε, τις διαδικασίες μετά τον πόλεμο και τις σχετικές αναφορές. Από ό,τι κατάλαβα και τα δύο μέρη, και η Γεωργία και η Ρωσία, έχουν ε, απευθύνει, ε, έχουν προσφύγει στο Διεθνές ε, Ποινικό Δικαστήριο για ξεχωριστούς λόγους. Θα ήθελα να ξέρω τι είδους συνέπειες θα έχουν αυτές οι συζητήσεις για το ποιος ήταν υπεύθυνο για τον πόλεμο αυτό και ποια ήταν ενδεχομένως κλίματα πολέμου κτλ. Και από ό,τι κατάλαβα το Δικαστήρια των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για πρώτη φορά αντιμετωπίζει ε, μία κατάσταση πολέμου. Νομίζω ότι έχουν γίνει χιλιάδες προσφυγές από πλευράς Γεωργίας. Και τέλος, για την έκθεση Ταλεαμπίνη, θα ήθελα να ακούσω δύο λόγια για το πώς ερμηνεύεται τα πορίσματά της. Η έκθεση αυτή θεωρώ δεν καταδεικνύει τίποτα. Το πόρισμα είναι ότι η κυρία Ταλιαβίνη δεν ε, μπόρεσε να διαπιστώσει μαζική κινητοποίηση των ρωσικών στρατευμάτων πριν από κάποια στιγμή. Τη ρώτησα λοιπόν, διαπιστώσατε ότι δεν υπήρξε τέτοια κινητοποίηση. Μας είπε όχι. Και αυτό αποτέλεσε βασικό πυλώνα των πορισμάτων της. Αν θα θέλατε λοιπόν να σχολιάσετε το θέμα αυτό. La parola a Έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Καταρχάς, για να επανέλθω στο ζήτημα της ε, εξασφάλιση της ε, συνεργασίας των διαφορών πλευρών στην περιφέρεια. Μου θυμίζει βέβαια αυτή η συζήτηση, οι συζητήσεις που είχαμε και τα τελευταία χρόνια, την εντύπωση δηλαδή ότι μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα μια μορφή περιφερειακής συνεργασίας για τις χώρες του Νότου Καυκάσου. Από την άλλη όμως υπάρχει δυνατότητα για συνεργασία και θα πρέπει να ε, επενδύσουμε σε αυτήν. και να προσπαθήσουμε να δούμε πόσο μπορούμε να ενθαρρύνουμε και να ενισχύσουμε μέσω του διαλόγου και των δυνατοτήτων των, της επικοινωνίας ίσως και της διαμεσολάβησης, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι εναλλακτική ως προς μια διαδικασία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω, όπως είπα και νωρίτερα, ότι είναι πολύ, πολύ, πολύ μακρινό στόχος η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τώρα το να κλείσουμε την πόρτα και να πούμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μεγάλο σφάλμα. Επίσης, τα Βαλκάνια βλέπω ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο παράδειγμα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η διαπεριφερειακή συνεργασία. Αλλά η διαφορά βέβαια είναι ότι στα Βαλκάνια υπήρχε η πρόπτικη ε, για την ένταξη και αυτό θα πρέπει να προσφερθεί και στον Κάφκασο. Οι τρεις χώρες ε, διαδραματίζουν ε, δαπανούν μεγάλο μέρος του ΑΕΠ τους στα στρατιωτικά, εξοπλισμού. εξοπλισμούς, με πρώτη τη Γεωργία 8% επί του ΑΕΠ το 2008, 3,2% η Αρμενία και 2,6% το Αζερβαϊτζάν. Δύο χώρες, τρεις χώρες φτωχές, αν το ξεχνάμε, που έχουν ανάγκη να αναπτύξουν τις οικοδομές τους, την παιδεία τους, την υγειονομική περίθαλψη και ε, ανταυτού σκορπούν τόσο μεγάλα ποσά στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς η χρήση της στρατιωτικής ε, ισχύω και βέβαια η εμπλοκή σε θερμή σύγκρουση είναι μια πραγματικότητα, μια, πιθανή, μια πραγματική πιθανότητα για τις χώρες αυτές. Για δε τις, ε, τα μαθήματα στα οποία αναφέρεστε ε, δεν έχω άμεση γνώση ότι όντως δίνουν τέτοια μαθήματα στα παιδιά, αλλά δεν το αμφισβητώ διότι είχαμε και στο παρελθόν στην, ε, Γεωργία τα στρατόπεδα, τα πατριωτικά στρατόπεδα όπως τα λέγανε, η πατριωτική κατασκήνωση και φαντάζομαι ότι μπορεί να συνεχίσει το ίδιο μέθοδος και τώρα. Για την UMM ε, φαντάζομαι ότι θα συνεχίσουν οι Ρώσοι να πιέζουν για να έχουν κάποιο σημείο πρόσβασης. Βεβαίως η UMM έχει κληθεί να συμβάλλει στον κοινό μηχανισμό στην Απχασία, θα πάει και στον Γκάλι και σε διάφορες συνεδριά, συνεδριάσεις ζήτησαν να προπάμε για να τους δώσουμε, να, μιλήσουμε και να ακούσουμε τα περί έναν κρατούμενο, φυλακισμένο δηλαδή νότιο το, ε, μπορούμε βέβαια να πάμε να τους ακούσουμε, να δούμε τι έχουν να πούνε, να δούνε και εκείνοι στην πραγματικότητα τι συμβαίνει. Από το 2008 είδαμε ότι σταμάτησαν αυτές οι αποστολές για λίγο. Θα, θα επανέλθουν όμως οι εκπρόσωποι του EUMM. για την Αρμενία και το ρόλο της ε, στην προσέγγιση. Ε, από τα όσα είπα ακούστηκε ότι κατηγορώ περισσότερο την Τουρκία γιατί νομίζω ότι η Τουρκία οπισθοδρόμησε, υπαναχώρησε σχέση με την αρχική της δέσμευση για την προσέγγιση με την Αρμενία τώρα και η Αρμενία σκληραίνει τη στάση της όπως επεσήμανε ο κύριος Βουλευτής και απειλεί να αποχωρήσει από τη διαδικασία που θα σήμερα ή να σταματήσει τη διαδικασία για την κύρωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει την πορεία αυτή η Αρμενία όμως εάν δει ότι από την Άγκυρα αποστέλλονται πιο θετικά μηνύματα γιατί εν τέλει τα χρειάζεται περισσότερο τα πρωτόκολλα αυτά η Αρμενία από τα χρειάζεται η Τουρκία. Άρα πιστεύω ότι θα συνεχίσει την πορεία της. Έστω και αν έχει σοβαρές εσωτερικές επιπτώσεις, πολιτικές επιπτώσεις η υπογραφή αυτών των πρωτοκόλων στο εθνικό επίπεδο και γι' αυτό είναι σημαντικό να βοηθήσουμε στη διαδικασία αυτή για να περιοριστεί ε, η ισχύ των εθνικιστικών δυνάμεων στην Αρμενία. Ευχαριστώ. Για τα όσα δεν κάλυψε η Σαμπίν, θα ήθελα να προσθέσω το εξή, ότι για τα οικονομικά ζητήματα, και μην με παρεξηγείτε, νομίζω ότι σωστά λέτε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ε, ευημερία, την ανάπτυξη και ότι αυτό πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις αντί να προσπαθούν ε, να διαιωνίζουν διαφορές. Θα έπρεπε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται και να οικοδομήσουν πάνω σε αυτές. Αλλά ε, θα σημειώσω εδώ ότι δεν αρκούν τα οικονομικά συμφέροντα για να λυθούν τα προβλήματα. Υπήρχε για ένα καιρό το επιχείρημα ότι εάν η γεωργία οικονομικά καταστεί ελκυστική, οι Απχάζοι και οι Νότιο Σετοί θα επέστρεφαν σε αυτήν. Όμως δεν αρκεί αυτή η οικονομική ελκυστικότητα, ε, η ε, έλξη, η ευρωστία οικονομική. Πρέπει και οι κυβερνήσεις να έχουν στάση η οποία να φέρνει κοντά τους πολίτες ε, των αποσχιστέντων εδαφών. Για τον Αγκόρνο Καραμπάχ τώρα θέλω να σημειώσω ότι είχε λησμονηθεί λίγο πολύ από το διεθνές ε, σκηνικό, από, τις, από τους διεθνείς παρατηρητές και τις αποστολές τους, πράγμα το οποίο βρίσκω λυπηρό γιατί ουσιαστικά έμεινε αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο, λησμονήθηκε και θα έπρεπε νομίζω να επανεκκινήσουμε τις επαφές μας, να τους δείξουμε ότι αναγνωρίζουμε το πρόβλημα και βέβαια το ότι έπαψε η Unomex στην ε, Απχασία, ότι δεν θέλουν οι Απχάζοι την ε, είναι, είναι λυπηρό, οι Απχάζοι δεν ε, ήθελαν να διώξουν την Ιουνομέκ, ήθελαν την παραμονή της και τη συνέχιση του ρόλου της. Αλλά δεν φαίνεται ότι είναι δυνατόν αυτό για το εγγύς μέλλον. Κάποια μέλη μεμονωμένα των προσωπιών πηγαίνουν και παρακολουθούν την κατάσταση και μάλιστα ορισμένοι από αυτούς γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση για την υπερδνηστερία αλλά και για την Απχασία και την Νότια Σετία. Θα ήθελα να πω ότι για την ε, Γεωργία είναι ιδιαίτερα μεγάλο το πρόβλημα γιατί οι κάτοικοι των δύο αυτών εδαφικών ε, των τρίτων έχουν ρωσική υπηκότητα και ω το πρόβλημα εξίσου σοβαρό για την Γεωργία όσο είναι και η υπερθνιστερία για τη Μολδαβία. Ε, Όμω οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να έχουν τη ρωσική υπηκότητα και μερικέ φορέ καλό θέλουν να κοιτάμε και τη δική του την οπτική, να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι λένε αντί να του καταδικάζουν αυτοί τις αποφάσεις λαμβάνουν για τους λόγους που θεωρούν ότι είναι προς το συμφέρον τους, για δικούς τους λόγους θεωρούν ότι είναι προς το συμφέρον τους και πρέπει να προσπαθούμε να τους καταλαβαίνουμε και όχι να ε, θεωρούμε δεδομένο ότι απλώς ε, λαμβάνουν κάποια απόφαση για να ενοχλήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από καπρίτσιο. Για την έκθεση θα ήθελα να σημειώσω ότι είναι μια και την ερώτηση της κυρίας Ταλιοδίνη. θα ήθελα να πω ότι η έκθεση είναι αρκετά περίπλοκη, δεν είναι εύκολο να ορίσουμε ε, υπετίους ε, ή να δούμε ποιος είναι εκείνος ο οποίος τράβηξε την ε, σκανδάλη. Κυρία Ταλτοβίνη, θα ήταν μάλλον σε δύσκολη κατάσταση αν επιδιώκαμε κάτι τέτοιο, ε, όπως και η ολόκληρη ομάδα της. Πάντως πρέπει να σημειώσουμε ότι τα θέματα της δικαιοσύνης και της ειρήνης είναι και περίπλοκα και αντικρουόμενα. Είδαμε ότι είχε προηγηθεί πριν από την παρουσία της εκεί ε, μια μεγάλη, μια έντονη αντιπαράθεση, ένας ε, χορός ε, επιθετικών στάσεων και δηλώσεων μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας που δεν ήταν δυνατόν να αποφύγουμε βέβαια αλλά το θέμα είναι πέραν αυτού τι μπορούμε να κάνουμε για να προχωρήσουμε και να αφήσουμε πίσω το παρελθόν τα κράτη έχουν τις ευθύνες τους και πιστεύω ότι η έκθεση καταγράφει αναλυτικά τις ευθύνες των δύο πλευρών και βέβαια είναι κατανοητό το γεγονός ότι θα πρέπει και ε, κάθε πλευρά να διασώσει τα προσχήματα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και ο καθένας να ε, αναλάβει τις ευθύνες του. Και αυτό, σε αυτό μπορούμε να τους βοηθήσουμε εμείς από τη διεθνή κοινότητα, μαζί με την ε, έννοια της ε, υποχρέωσης λογοδοσίας για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλαμ, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές ιδιαίτερα την κυρία Φίσερ που μας ε, παρουσίασε τις επιτυχίες, τις αποτυχίες και τα εμπόδια το οποίο και καταδεικνύει ότι οι αποτυχίες και τα εμπόδια είναι τα πιο πολλά. Και συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο Σέμπαριν και με άλλους συναδέλφους ότι η χρήση, η συνεχιζόμενη χρήση του όρου παγωμένων σειράξεων έχει πλέον ξεπεραστεί και είναι και παραπλανητική αν θέλετε. Η Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας, η Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Κοινοβουλίου μίλησε πέρσι και παρουσίασε μια έκθεση για τις μετασοβιωτικές αυτές συγκρούσεις και με αυτό το απικιο κρατικό παρελθόν δεν θέλω να δαιμονοποιήσω την Ρωσία αλλά θα πρέπει πιστεύω να αντιμετωπίσουμε τις πραγματικότητες. Για παράδειγμα, τις ε, δράσεις της Ρωσίας που ξεκίνησαν το 1992 για να καθιερωθεί η ρωσική επιρροή, οι οποίες κινούνται, κινούνται κατά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσφέρουμε στις χώρες, τα έθνη της περιοχής αυτής, μία ευκαιρία για να αποφασίσουν μόνες τους να ταχθούν υπέρ της δημοκρατίας, της οικονομικής ανάπτυξης και δυστυχώς το ρωσικό μοντέλο δεν προσφέρει πολύ απλά τα στοιχεία αυτά. κοιτώντα την απόλυτη αποτυχία της ρωσικής πολιτικής για την ε, καταστολή στην ε, Τσετσενία, είναι σαφές ότι δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Θα πρέπει να είναι έντονη η παρουσία μας θα συμφωνούσατε με δύο συμπεράσματα. Καταρχάς, ότι τα ρωσικά στρατεύματα που ε, έχουν ε, το ρόλο διεθνών ειρηνευτικών δυνάμεων δεν μπορούν να θεωρηθούν ως τέτοια πλέον, γιατί έχουν χάσει το καθεστώς αυτό. Και αυτό θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Και κατά δεύτερον, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται και θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το βάρος της για να κάνει την Ρωσία να τηρήσει τις δεσμεύσεις του Σεπτεμβρίου του 2008. Γιατί δεν έχει νόημα να αναπτυχθούν επαφές με τις διάφορες αυτές οντότητες χωρίς πρώτα η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει δυνατότητα να αποστείλει ε, αποστολές παρατηρητών στην Νότια Απχαζία και στην ε, Οσουτία. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Κυρίλοφ, ο οποίος θα παρουσιάσει και το κείμενό του λίγο αργότερα, ότι η αντίδραση, η απλή αντίδραση στα τεκτενόμενα και στις κρίσεις δεν θα αποτελέσει στο μέλλον μία βιώσιμη λύση. Θα πρέπει να υπάρξει δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Δημοκρατία και προς την πολιτική της Ένωσης. Και τελευταία ερώτηση. Τι πιστεύετε. αναφορικά με την διστακτική στάση της Ένωσης απέναντι στις ε, παραβιάσεις της Ρωσίας και τις ε, επιδρομές της ε, στη Γεωργία θα μπορούσαν να, ενθαρρύνουν, να ενθαρρύνει αυτή η στάση της Ένωσης στη Ρωσία για παρόμοιες δράσεις και στη Μολδαβία και αλλού. Ο κύριος Λίζεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Δόκτωρ Φίσερ μας είπε, ή Δόκτωρ, συγγνώμη, μας είπε πως ε, υπήρχε ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση των ΗΠΑ στον ε, Νότιο Κάφκασο και από τότε που έχουμε την αλλαγή κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον. Αυτό είναι σωστό, το τον μάλλον καθώς είχα την ευκαιρία στο Χάλιφαξ σε ένα συνέδριο να συναντήσω και να συζητήσω με Αμερικανούς πολιτικούς και είπαν ότι σε άλλες θερμές περιοχές του κόσμου όπως Αφγανιστάν, εκεί Ανατολή κλπ. χρειαζόταν να υπάρξει μια πολύ στενή συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την... Ε, Στι Αλλά σε ό,τι αφορά τον Νότιο Κάφκασο και άλλες ε, παρόμοιες περιοχές, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την επίλυση αυτών των σειράξεων, να αναλάβει ένα πιο ενεργό ρόλο. Τι πιστεύετε σχετικά με τις δηλώσεις αυτές των Αμερικανών πολιτικών. Παρατηρήσατε κι εσείς μια μείωση του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για να φέρουμε και για δραστηριότητε πολιτικού, διπλωματικού και οικονομικού χαρακτήρα για ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών. Ευχαριστώ. Απάντηση παρακαλώ. Να ξεκινήσω με μερικά σύντομα σχόλια. Τώρα για να χρησιμοποιήσει πίεση και επιρροή η Ευρωπαϊκή Ένωση προ τη Ρωσία προκειμένου να σεβαστεί τις δεσμεύσει τη, αυτό ναι είναι γεγονό. Ταυτόχρονα όμω, γνωρίζουμε πω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει και τόσο πολύ επιρροή στην Σοβιετική Ένωση και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Εντάξει, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το βάρος μας, την επιρροή μας, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει ποιες είναι οι πραγματικότητες επιτόπου στις περιοχές και να αναπτύξει κάποιες συγκεκριμένες και εκλεπτισμένες πολιτικές όχι απέναντι στη Ρωσία, αλλά αναλύοντας ε, προσεκτικά τα, το τι συμβαίνει επί τόπου. Θεωρούμε πως ε, η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει πάρμες ε, πρακτικές στην Κρυμαία και στην Μολδαβία. Ο Τζόναθαν κάτι είπε σχετικά με την υπερδνηστερία. Νομίζω πως η κατάσταση στην υπερδνηστερία είναι πολύ λιγότερο εκρηκτική και διαφέρει σημαντικά από την κατάσταση στην Γεωργία, Νότιο Οσετία και Απχαζία. Ναι, εκεί μπορεί να υπάρξει στρατιωτική κλιμάκωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ε, ανησυχούμε για την παρουσία των ε, ειρηνευτικών στρατευμάτων της Ρωσίας στην υπερνηστερία. Αυτό είναι προβληματικό, πρέπει να το έχουμε κατά και να το παρακολουθούμε. Τώρα η κατάσταση στην Κρυμαία και πάλι ε, είναι πολύ διαφορετική. Και εδώ θεωρώ ότι είναι απίθανο η Ρωσία να ε, προβεί σε χρήση στρατιωτικής ε, δύναμης ε, διότι αυτό θα έχει πολύ πιο σημαντικές επιπτώσεις για την Ρωσία. Και η Ρωσία μπορεί να περιμένει κάποια πλεονεκτήματα από τις προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία. Δεν νομίζω ότι η Ρωσία προβλέπει μια ε, στρατιωτική επέμβαση σχέση με την Ουκρανία θα ε, ακολουθήσουν μια διαφορετική πορεία μετά από τις προεδρικές εκλογές και αυτό το γνωρίζει η Ρωσία. Ευχαριστώ. σχολιάσω και, και εγώ κάτι γιατί μιλήσατε για τη Ρωσία ως μοντέλο και για τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτό, συμφωνώ. Αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι μπορεί να έχουμε εμεί τεράστια προβλήματα με την ρωσική δημοκρατία. Ας πούμε, ο λαός της Απχαζίας δεν έχει άλλη επιλογή παρά μόνο μία πιο στενή σχέση με τη Ρωσία και αυτό αφορά την ε, απορρόφηση της Απχαζίας από τη Ρωσία. Αν δεν κοιτάξουμε λοιπόν και δεν συμμετέχουμε πιο ενεργά, αν δεν σπάσουμε αυτόν τον κύκλο απομόνωσης, θα συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτόν τον φαύλο κύκλο. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πρόσβαση, λέτε, δεν θα πρέπει να συμμετέχει. Νομίζω ότι αυτό αντιστρέφει τη σειρά των επιχειρημάτων. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συμμετέχουμε, πρέπει να συμμετέχουμε ακριβώς επειδή δεν έχουμε πρόσβαση για να έχουμε μία σχέση σε διαφορετικούς, με διαφορετικούς όρους στο μέλλον, λέγοντας ε, ότι δεν έχουμε πρόσβαση και άρα δεν θα συμμετέχουμε, δεν θα δραστηριοποιηθούμε, νομίζω ότι γράφουμε ήδη τη μοίρα μας. Ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο Κύριε Λόφου που θα μας παρουσιάσει την έκθεσή του σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Κάφκασο. Θα μαζέψουμε ερωτήσεις, θα τις ομαδοποιήσουμε και θα προχωρήσουμε. Συνάλφε Κύριλοφ, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ε, προσκεκλημένους μας για όλες τις καλές ιδέες που ακούσαμε θα πρέπει να πούμε ότι ο πόλεμος μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας καταδεικνύει πόσο ευάλωτη είναι η γειτονία προς Ανατολάς και πόσο σημαντικές είναι αυτές οι σειράξεις για την περιοχή και τη σταθερότητά της και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δραματίσει νέο ρόλο συμμετοχής για την μεταρρυθμίση, για τη ε, μόρφωση της ε, περιοχής σε μια περιοχή σταθερότητας. Μετά από τον πόλεμο η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέδειξε ότι έχει την δυνατότητα να κάνει να διαδραματίσει τον ρόλο αυτό. Και η θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και η δημιουργία της θέσης της ύπατης εκπροσώπου καταδεικνύουν ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άμεση γειτονία. Για να μην ξεχνάμε ότι πολλές χώρες μέλη της Ένωσης έχουν σύνορα με τη Γεωργία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποτυπωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο α, οι καταστάσεις και οι δυναμικές που επικρατούν στην περιοχή. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Κόεν, ο οποίος μιλάει για μία πιο μεγάλη πολιτική ικανότητα, η οποία είναι πολύ σημαντική, θεωρώ. Δεν μπορούμε απλά να μένουμε μέτοχοι και να παρακολουθούμε τι συμβαίνει στην περιοχή. Και αυτό αφορά και τις σειράξεις. Επέλεξα να ξεκινήσω με θέματα ασφάλειας, γιατί θεωρώ ότι πρόκειται για τα ορόσημα για την επιτευξή σταθερότητα στην περιοχή. γιατί η κατάσταση των ανεπίλητων διαφορών μπορεί να προκαλέσει κατάχρηση της κατάστασης, όταν είπε ο κύριος Κοέν επίση ότι το Ναμπόρνο Καραμπάχ έχει βγει από το ραντάρ. Για να τα πούμε τα πράγματα ευθέως, η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνεται γι' αυτό. Και γι' αυτό ζητάω στην έκθεση πιο ενεργό ρόλο της Ένωσης. Μιλάω για την ευρωπαϊκή εντολή και για άλλα θέματα, τα οποία μπορεί να φαίνονται πολύ φιλόδοξα, αλλά θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψη των συναδέλφων. Επίσης, ε, τονίζω τις ε, επαφές μεταξύ των λαών και όλα τα μέτρα οικοδόμησης ε, εμπιστοσύνη που μπορεί να προάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει κάποιες πολύ καλές ιδέες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαι σίγουρος ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι όροι για να διαδραματίσει το ρόλο της εκεί η Ένωση. Η Ένωση ασκεί την ήπια δύναμή της ήδη και με την πρωτοβουλία ανατολικής εταιρικής και σχέσης που στην τελική ανάλυση θα προσεγγίσει τις χώρες αυτές προς την Ένωση. Αυτή η διαδικασία προσέγγισης θα σταθεροποιήσει την περιοχή και θα πρέπει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει την διαδικασία αυτή. Και σημαντικό είναι το καθεστώς για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων. Και το συμπέρασμα των ε, συμφωνιών εμπορικών σχέσεων που θα βελτιώσουν τις ε, σχέσεις και το οικονομικό κλίμα στις χώρες. Επίσης, ε, τόνισε τη σημασία του φόρουμου των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και της ε, βελτίωση των σχέσεων των χωρών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης σκοπεύω να εστιαστώ στην οικοδόμηση των θεσμών που προσφέρει η εταιρική σχέση προς Ανατολάς για να βοηθήσει τις χώρες αυτές να επωφεληθούν από τις πρωτοβουλίες μας. Το δεύτερο τμήμα της έκθεσης εστιάζεται στις προσπάθειες των χωρών αυτών για τον εκδημοκρατισμό, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου. Θα πρέπει να γίνονται απόλυτα σεβαστές αυτές οι αρχές. Και αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που έχουν ήδη γίνουν, θα πρέπει να γίνουν όμως πιο πολλές προσπάθειες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία των δικαστικών και το καθεξής. Στο τρίτο τμήμα της έκθεσης εστιάζομαι σε οικονομικά θέματα και την κοινωνική ανάπτυξη. Είναι σημαντική η όρη αυτή για την επίτευξη της σταθερότητας στην ε, περιοχή και φυσικά όπως είπαν και οι συνάδελφοι, αυτό θα είχε μεγάλη επιρροή και για τους πολίτες στις χώρες αυτές. Να μην ξεχνάμε ότι απέχουν οι περιοχές αυτές μόνο 15 χιλιόμετρα από τον ε, αγωγό του Μπακού. Και θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες και για την ενεργειακή ασφάλεια που θα διασφαλίσει και τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Και να μην ξεχνάμε ότι θα αρχίσουν οι ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία, αλλά σημαντική στο σημείο αυτό είναι και η Κίνα. Και ότι επίσης μεγάλο τμήμα του φυσικού αερίου ρέει από το Τουρκμενιστάν προς την Κίνα μιλάμε για διάφορα προγράμματα υπάρχουν τόσα πολλά έργα, αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι χωρίς πολιτική παρουσία πολύ απλά θα μείνουμε απλοί, απλή ε, απλοί παρατηρητές στην όλη διαδικασία. Να πω επίσης ότι η Ρωσία πληρώνει καλές ε, τιμές για, τα, για το αέριο αυτό. Είναι καλύτερες τιμές από, ότι, από αυτές που πληρώνει η Τουρκία. Θα πρέπει λοιπόν να συμμετάσχει πιο έντονα η Ευρωπαϊκή Ένωση και να, σε ό,τι αφορά τα θέματα ενέργεια στην περιοχή και να εξασφαλίσει μια πιο διαφοροποιημένη προμήθεια ενεργειακή στην Ένωση. Σταματάω εδώ και θα ήθελα να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων. Και ελπίζω η έκθεση αυτή να κάνει πιο σαφή το ρόλο της Ένωσης στην περιοχή. Bene, grazie collega Ευχαριστούμε συνάδελφε Κύριλοφ. Θα ήθελα να λάβω το λόγο διότι με, εντυπωσίασε μια δήλωση που έκαναν οι συγητές σχετικά με την κατάσταση των Ογκόρνο Καραμπάχα. Η δήλωση λέει ότι Αρμενία και Αζερβαϊτζάν δεν ενδιαφέρονται για μεγαλύτερη εμπλοκή συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ πως αυτό είναι ιδιαίτερα ενδεικτικό το, σε ό,τι αφορά το γόητρο, το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι επιθυμούμε να υπάρξει μεγαλύτερη εμπλοκή, συμμετοχή στην κατάσταση των Αγκόρνη Καραμπάχ αλλά και στην περιοχή ευρύτερα, αλλά αυτή η συμμετοχή δεν μπορεί να είναι άμεση και να γίνει μέσω κάποιας χώρας μέλους Σύμφωνα με το ΜΕΣΚ η Ευρώπη αποκλείεται, είναι παρούσα η Γαλλία, αλλά δεν έχει λάβει ούτε καν εντολή από πλευράς Ευρώπης. Άρα δρά αποκλειστικά για λογαριασμό της. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω πώς η Ευρώπη μπορεί να συμμετάσχει και να αποκτήσει πολιτικό κύρος και όχι μόνο να παρέχει βοήθεια στους πρόσφυγες και να συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών. Και κάτι ακόμα που αφορά στον παρουσίαση του, του ψηφίσματος να συγχαρώ τον συνάδελφο που συμφωνώ απόλυτα με τα λεγόμενά του, ειδικά τον ρόλο που μπορεί να έχει αυτή η εταιρική ανατολική σχέση που σε σχέση με την δήλωση της Πράγας προβλέπει παρεμβάσει διαφόρων, διαφόρων μορφής δημοκρατικού, κοινωνικού, πολιτικού, σταθερότητας ε, και ασφάλειας, ε, αλλά και ασφάλειας στην, ε, στην στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι φορά την ασφάλεια της Γεωργίας, εάν η άλλη πλευρά, η εμπλεκόμενη πλευρά ε, είναι η Ρωσία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανατολική συμφωνία. Υπάρχουν δύο ακόμα εμπλακόμενα μέρη που είναι το Αζερμπαϊτζάν και η Γεωργία που είναι άμεσα ενδιαφέρον, διότι η διευθέτηση αυτής της εμπλοκής, σημαίνει και την μεγαλύτερη ή μικρότερη συμμετοχή μας ε, στην διευθέτηση του προβλήματος. Ρωτάω λοιπόν τον συνάδελφο Κύριλοφ, η ειρήνευση και η επίλυση του ε, προβλήματος του Ναγκόρνη Καραμπάθ είναι ε, και οι σχέσεις με, με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν θα ήταν μία προϋπόθεση προκειμένου να εγγυηθούμε την ε, επιτυχία αυτής της ε, εταιρικής ανατολικής σχέσης. Ο κύριος Μπιζάντζουτς έχει το λόγο. Συγγνώμη για τη φρικτή μου προφορά. Κύριε. Αλλά Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι πρέπει να προφέρετε το όνομά σας, κυρία μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έξι χρόνια είμαι στο Ε. Θα μπορούσε κάποιος να μάθει το όνομά μου, αλλά έχω συνηθίσει να το προφέρουν ανάποδα. Από το Μαυροβούνιο είναι το όνομά μου, ε, ωστόσο έχω γεννηθεί στη Βοσνία και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει και σύγκρουση και τι σημαίνει και προσφυγιά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα τις συζητήσεις. Έχω μια σειρά σχολείων και εγώ να προσφέρω. Αλλά, μια και δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα περιοριστώ σε κάποιες σύντομες ε, δηλώσεις ε, στα όσα είπε ο κύριος Κύριλοφ, γιατί είμαι σχεδόν για την έκθεση από πλευρά του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κύριλοφ. Ήταν καλό το κείμενο ως βάση για τις εργασίες μας. Ασφαλώς θα κάνω μια-δύο τροπολογίε κι εγώ, αλλά πάνω απ' όλα δεν θέλω να ευχαριστήσω την υποστήριστή μου προς τον κύριο Κύριλοφ για την αναγκαιότητα μια κοινή στρατηγική, την οποία θεωρώ και εγώ απαραίτητη. Όπως είπα, έχω προσωπική εμπειρία από όλα αυτά και έχω προσωπική εμπειρία από το γεγονό ότι όταν δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στραφή στρατηγική, οι συγκρούσει, γίνονται αναπόφευκτες ή καταλήγουν ανεπίλητες. Όταν έχουμε στρατηγική καταφέρνουμε καλά αποτελέσματα. Με την ταχαία παρέμβαση παραδείγματα στην Ουκρανία, τη Γεωργία και αλλαχού. Επίση, η σημασία τη οικονομική ε, συνεργασία και τη παρουσία τη κοινωνία των πολιτών ω σταθεροποιητικού παράγοντα θα πρέπει να υποβαθμιστεί. Είναι πολύ σημαντική. Θα ήθελα και εγώ να καταθέσω κάποιε θετικέ τροπολογίε. Και τώρα επιτρέψτε να περάσω σε ένα κάπω πιο κρίσιμο σημείο, κάπω πιο επικριτικέ παρατηρήσει προ την ελευθερία ε, των μέσων μαζική ενημέρωση και τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, τη ε, πολιτικής ελευθερία ιδιαίτερως, που θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερα όσον αφορά το Αζερβαϊτζάν και από την ε, ανακοίνωση και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την έκθεση μάλλον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είδαμε σήμερα, βλέπουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ επικριτική απέναντι στην κατάσταση αυτή. Βλέπω ότι ο κύριο Κυρίλοφ δεν είναι το ίδιο επικριτικό απέναντι στο πρόβλημα και θα ήθελα να καταθέσω τι σχετικέ τροπολογίε. Αλλά μακάρι να έχουμε την ευκαιρία να ξανασυστήσουμε την έκθεση αυτή, γιατί έχουμε πολλά ακόμα πράγματα να πούμε. Άλλο παραβάσει παρακαλώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω τόσο είπε η κυρία Έντρι Ω Τσικ. Ως την ε, θέση του ΕΛΚ για την έκθεση Κυρίλοφ, για την οποία και εγώ τον συγχαίρω. Ε, φρονώ ωστόσο ότι ορισμένα πραγματικά περιστατικά που καταγράφει η έκθεση δεν είναι επαρκή. γιατί όχι μόνο έχουμε εσωτερικά εκτοπισμένους, αλλά και πρόσφυγες. Αρμένοι χρειάστηκε να φύγουν από το Αζερβαϊτζάν, να, με, θα τοπιστούν στην Αρμενία. Ε, είχαμε επίσης βία επεισόδια μετά τις εκλογές που δεν καταγράφονται πιστά στο κείμενο. Ο κύριος Νικόλ Πασινιανέ ναι, είναι δημοσιογράφος, αλλά αυτό που έχει κάνει και ο λόγος για τον οποίο έχει ασκηθεί εναντίον του δίωξη δεν είναι ε, δεν έχει να κάνει με την εκτέλεση των δημοσιογραφικών του καθηκόντων ή εργασιών, αλλά με τις πολιτικές του τοποθετήσεις. Ως πολιτικός διώκεται. Και αυτά θα ήθελα να τα διορθώσουμε με τις τροπολογίες. Αλλιώς η έκθεση είναι πολύ καλή. Κύριε Νέιτς, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη από τους εμπεριογνώμονες γιατί δεν άκουσα όλες σας τις παρουσιάσεις. Τις ε, διάβασα ωστόσο. Ακούγοντας τι λένε οι συνάδελφοι, μου κάνει εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχει μία αντίφαση ή μία επιπλέον δυσκολία η οποία ανακύπτει από το ότι πιστεύουμε ότι εμείς ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε δικαίωμα να προβάλλουμε τεράστιες απαιτήσει έναντι χωρών οι οποίες βρίσκονται εν το μέσο σειράξεων για να βελτιώσουν την κατάστασή τους, για να εναρμονιστούν με τις αξίες που θεωρούμε ορθές και εκ παραλλήλου δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε να επιλύσουν τις σειράξεις αυτές. Και ακούγοντας αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, αναρωτιέμαι σε ποιο βαθμό Αυτές ε, οι παράλληλες στάσεις μπορούν να συμφιλειωθούν. Θέλουμε από τον Αζερμπαϊτζάν να κάνει κάτι για την σύραξη, αλλά παράλληλα ζητάμε ορθώς να βελτιωθεί ο δημοκρατικός χαρακτήρας, να υπάρχει ελευθερία τύπου, να μην υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι σωστά και δίκαια. Το θέμα όμως είναι κατά πόσο πρόκειται για μια στάση που θα ενθαρρύνει το Αζερβαϊτζάν τελικά ή και άλλα κράτη φυσικά. Και θα το βοηθήσει να επιλύσει την ε, σύγκρουση. Τι είναι η προτεραιότητά μας, ποια είναι η προτεραιότητά μας, να το θέσω έτσι. Ποια είναι η προτεραιότητά μας, να δούμε όλες οι χώρες αυτές να συμμορφώνονται με τις αξίες μας ή να λυθούν πρώτα οι συγκρούσεις ή και τα δύο ταυτόχρονα και ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση για να το πετύχουμε αυτό. Εγώ έχω την εντύπωση ότι σε κάθε περίπτωση η απομόνωση μιας χώρας ή ενός λαού σίγουρα δεν αποτελεί λύση. Το έχουμε δοκιμάσει σε διάφορα μέρη, στον Νότιο Κάφκασο, σε άλλα γειτονικά κράτη και πολύ απλά δεν έχει λειτουργήσει αυτό ως προσέγγιση. Άρα, ναι, θα πρέπει να συμμετάσχουμε, αλλά πώς. Θα προσπαθήσω να διατυπώσω πιο συγκεκριμένα τις απόψεις μου όταν θα έχω διαβάσει και την έκθεση του κυρίου Κυρίλοφ για να υποβάλλω τροπολογίες, αλλά επειδή ήμουν υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στη χώρα μου μεταξύ του 2000 και του 2003, και μου κάνει την εντύπωση, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι κάθε προεδρία εκπεριτροπής στην Ένωση προσπαθεί, καταβάλει προσπάθειες για να βελτιώσει την κατάσταση και μετά δεν τα καταφέρνει, τι να γίνει, το προσπαθεί η επόμενη Προεδρία. Η πολιτική αυτή δεν χαρακτηρίζεται από συνέχεια και συνέπεια. Προσπαθούμε μία, ε, να εφαρμόσουμε ένα μέτρο, μετά κάποιο άλλο μέτρο. Δεν υπάρχει συνοχή και δεν υπάρχει μια βαθιά κατανόηση της περιπλοκότητας και της μοναδικότητας των καταστάσεων αυτών. Ο συνάδελφος Μιρσκι. Γεια σας, συνάδελφοι. Διάβασα το σχέδιο έκθεσή σας και θα ήθελα διευκρινήσεις. Στο πέμπτο σημείο μιλάτε για προνομιούχους, προνομιακούς, ε, ε, προνομιακά μέρη σε ό,τι αφορά τις συγκρούσεις αυτές. Ποιος εννοείται, τη Ρωσία, αν τη Ρωσία εννοείται, γράψτε Ρωσία. Στο άρθρο 12 μιλάτε για εθνική κάθαρση, κάθαρση για την Γεωργία μιλάτε ή για την Απχαζία. Θέλω πιο συγκεκριμένα στοιχεία να μας, να μας δώσετε. Γιατί και εγώ έχω πάει στην ε, Οσοτία, όπου ο στρατός της Γεωργίας έχει σκοτώσει χίλιους και πλέον Απχαζούς. Ποιους εννοείται λοιπόν, κύριε Κυρίλοφ. Θα πρέπει να δώσετε συγκεκριμένα στοιχεία στην έκθεσή σας. Ultimo intervento mm, del collega Kelam che riinterviene, immagino per una precisazione. Θέλετε να λάβετε λόγο διευκρίνηση φαντάζομαι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατανοώ τις ανησυχίες ε, της συναδέλφου Νέιτ. Πρέπει να είμαστε συνεκτικοί και να αποφύγουμε να επιβάλλουμε τα πρότυπά μας σε κυρίαρχα κράτη. Αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα να μας υπενθυμίσω ότι αυτά τα τρία κράτη έγιναν μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ιδία θελήση και έχουν αναλάβει δημοκρατικές δεσμεύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε να συμπεριφέρονται με βάση αυτές τις δημοκρατικές αξίες. Ευχαριστώ. Allora, la replica al collega Λοιπόν, ο κύριος Κύριλοφ και μετά ε, μερικά λόγια από τους ε, εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσουμε με τα δικά σας σχόλια φυσικά. Αναφερθήκατε στο ζήτημα της ε, εντολής ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Η ομάδα του Μίνσκ είναι ε, σε αυτήν την ομάδα συμμετέχουν πολλά φιλοευρωπαϊκά κράτη αλλά Έχοντας και την συνθήκη Λισαβόνας που ετέθηκε σε ισχύ, χρειάζεται να βρούμε κάποιον μηχανισμό ώστε να δούμε τους σύνεγγες στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, διότι μερικές φορές η Κομισιόν λαμβάνει αλληλογροθοκοπούμενες εκθέσεις. η Γαλλία αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο πολύ πιο στεναρό. Αυτό εννοούσα. Εντάξει, είναι κάτι που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, να ακούσουμε τις απόψεις των συναδέλφων, αλλά είναι παράδοξο εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να μην γνωρίζουμε τίποτα και να μην λέμε τίποτα για τα τεκτενόμενα στην ομάδα Μίνσκ. Και αυτό ενδεχόμενα είναι ο λόγος για τον οποίο εδώ και τόσο καιρό αυτή η διαδικασία παρατείνεται, παρατείνεται χωρίς να αποδίδει. Τώρα για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Πιστεύω πως πρέπει να υπάρχει συμμετοχή της Ρωσίας. Εξάλλου πιστεύω ότι έχει ήδη ξεκινήσει αυτή η εμπλοκή της. Ακούσαμε τη δήλωση της Μόσχας. Έγινε μια συνάντηση στο Σότσι τις τελευταίες μέρες. Η Ρωσία έχει πολύ ισχυρή παρουσία στην Αρμενία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί, τουλάχιστον σε ό,τι φορά τον Αγκόρνη Καραμπάχ. Ελπίζω να μην προκαλέσουμε κάποια ένταση με δυνάμει κάποιον ισχυρότερο ρόλο που θα διαμαρτύρει η Ρωσία, αυτό δεν το επιθυμούμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ξεανάμιξη της Ρωσίας. Αλλά και υπάρχει συμμετοχή και της Τουρκίας. Κυρία Ιμπρεζάζιτς, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θα κοιτάξω ξανά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά εδώ έχει το ζήτημά με σχέση με τα όσα είπε η κυρία Νάιτς. Ναι, θα πρέπει να έχουμε την εντολή μας και να ενθαρρύνουμε τα κράτη της περιοχής χωρίς ε, να έχουμε κάποιες υπερβολικές προσδοκίες, διότι αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι να πετύχουμε πρόοδο. Γι' αυτό και εγώ θέλω να προωθήσω τον πολιτικό ρόλο που μπορούμε να διαδραματίσουμε, διότι θεωρώ πως ε, αν υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία μας, τότε μπορούμε να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση και σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και σε θέματα εκδημοκρατισμού. Αν ε, πρέπει να δούμε από αυτή την πλευρά την διαδικασία. Διότι αν δεν μπορείτε να ασκήσετε πίεση ή επιρροή, τότε εντάξει. Παραμένουμε στα λόγια και στους ευσεβείς πόθους. Ε, το το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και οι εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από το όργανο αυτό θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν. Χρειάζεται λοιπόν μια ισορροπία εδώ. Όπως γνωρίζετε πριν από την πρωτοχρονιά ψηφίσαμε τις εκθέσεις για την πρόοδο και εγώ τότε είχα την εντύπωση πως ε, τα άτομα αυτά θα απελευθέρονταν. Απελευθερώνονταν. 99 άτομα απελευθερώθησαν αλλά οι δύο bloggers παραμένουν στη φυλακή. Πρέπει να παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις <coughs> και γι' αυτό αναφέρω εδώ τους δύο bloggers στο ψήφισμά μου. Γιατί αυτοί συνεχίζουν να παραμείνουν στη φυλακή. Τώρα, παρατήρηση του κυρίου Κασουλίδη. Συμφωνώ με το ζήτημα των προσφύγων και το υποστηρίζω. Τώρα, σε ό,τι φορά τα, κάποια βία γεγονότα, μερικές φορές ε, αυτά συμβαίνουν, το ξέρουμε πολύ καλά ως Κοινοβούλιο. Τώρα, κύριε Σπίρσκι, πιστεύω ότι είναι σαφές. ναι φυσικά ανέφερα την Νότιο Σετία και την Αυχαζία. Και καταλαβαίνετε ότι το ενδιαφέρον μου είναι ξεκάθαρο. Θα περιμένουμε τις τροπολογίες σας. Α, το ζήτημα επίσης της εθνοκάθαρσης. Δεν μπορούμε να το ανεχτούμε, το θεωρούμε παράδεκτο και φυσικά αν έχετε τροπολογίες ευχαριστώ να τις συζητήσουμε. Αλλά και εδώ το κείμενό μου θεωρώ ότι είναι σαφές. Ευχαριστώ. Μια γρήγορη παρέμβαση. Τελική παρακαλώ. Πρόεδρε, συγγνώμη, θα ήθελα όμω να απαντήσω στην ερώτηση σα ω προ το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον Αγκόρνο Καραμπάχ, έτσι ώστε να υπάρξει παρεξήγηση, να προέκυψε παρεξήγηση προ αυτά που είπα. Δεν είπα ότι περιμένουν οι Αρμένοι την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αγκορνο Καραμπάχ. Δυστυχώς θα μπορούσε να δραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικό ρόλο στον Αγκόρνο Καραμπάχ και πριν και μετά τη διευθέτηση της διαφοράς και σε στρατιωτικό και σε πολιτικό επίπεδο και ω προς την υποβοήθηση των εκτοπιστέντων ε, να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Πλην όμως το στάδιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επαρκή αξιοπιστία σε επίπεδο Αζερών, Αζέρων ή Αρμενίων για να δραματίσει τέτοιο ρόλο. Δεν έχουμε πάει εκεί, ούτε στις περιοχές, ούτε έχουμε και κάνει τίποτα για τους εκτοπιστέντες που βρίσκονται στο Αζερβαϊτζάν αυτή τη στιγμή κατεστημένοι. Άρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει πως αξιοπιστία και εμπιστοσύνη από πλευρά των Αζέρων και των Αρμενίων για να μπορέσει μετά να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην ε, διαφορά αυτή μέχρι ότου διευθυντηθεί και ελπίζουμε και αφού διευθυντηθεί. Ευχαριστώ. Κλείνοντας, δεν ήθελα να πω, να υπενθυμίσω την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών που μετατίθεται στις 17 Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Για όποιον ενδιαφέρεται. 17 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ πολύ τους προσκεκλημένους μας. Ένα μικρό διάλειμμα για να περάσουμε μετά στην ε, συζήτηση του μηχανισμού ΕΝΠΗ Ανατολή, ένα στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση τη Ανατολική Ανατολική Σχέση για την περίοδο 2010-2013, ανταλλαγή απόψε με την Επιτροπή. Bene, colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Stamane c'è stata. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Σήμερα κάναμε μια συζήτηση για την ε, για το θέμα της γειτονίας ε, του Νότου και τώρα θα ζητήσουμε το ζήτημα της γειτονίας προς Ανατολές. Κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων πρέπει να δίνουμε κάποιους πολιτικούς προσανατολισμούς σχετικά με το έργο της Κομισιόν. Οι εκλογές μας ε, από μας ε, προσδοκούν όχι μόνο την καλή χρήση των κοινοτικών κονδυλίων αλλά και την χρησιμοποίησή τους ε, με βάση τις προτεραιότητες της κοινή εξωτερικής μας πολιτικές. Η Κομισιόν προτίθεται να εγκρίνει τις νέες στρατηγικές προτεραιότητες ε, που διαπραγματεύεται με τις ε, δικαιούχες χώρες για το 2011-2013. Και στο σημείο αυτό χρειάζεται να παρέμβει η Κομισιόν μας, η Επιτροπή μας. Ε, έχουμε κάποιες ε, αναλύσεις ε, από πλευράς κομισιών, κάτι που θα μας βοηθήσει στην συζήτηση. Η διάσκεψη της Πράγας το Μάιο 2009 για την σύσταση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το 2009 η Κομισιόν ξεκίνησε την αναθεώρηση της χρηματοδοτικής αρρωγής που χορηγείται στις χώρες γειτονίες που μπλέκονται σε αυτή την εταιρική σχέση. Να δώσω το λόγο τον κύριο Τζον Κίαρ, υπεύθυνο για την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τον Νότιο Κάφκασο στην ε, Γενική Διεύθυνση Ρέλεξ, ώστε να μας παρουσιάσει εν συντομία τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση στο πλαίσιο της αναθεώρησης και δει στο ζήτημα της ερετίκης προσέγγισης αυτής της περιοχής από σήμερα μέχρι το 2013. Παρακαλώ. Thank you very much. Uh, distinguished... Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμο μέλη του Κοινοβουλίου. Με μεγάλη χαρά έρχομαι να προσφέρω τις απόψεις μου από τις δικές σας για την ευρωπαϊκή ε, στρατηγική για την ανατολική εταιρική σχέση με τους ανατολικούς μας εταίρους και τη Ρωσία, το ENPI όπως το ονομάζουμε. Και θα ήθελα ξεκινώντα να πω μερικά λόγια για το στόχο, τις βασικές, τα βασικά συμπεράσματα και το πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης και σύντομα στη συνέχεια θα ε, αναφερθώ στις χώρες μεμονωμένα και βεβαίως θα είμαι σε θέση σας μετά για όποιες ερωτήσεις έχετε ενδεχομένω. Θα θυμάστε ενδεχομένω ότι Στόχο τη ενδιαμέσης αναθεώρηση είναι να εξετάσει με στρατηγικό πνεύμα την ε, κατάσταση στι χώρε ENPI, τι ανατολικέ χώρε ENPI και τι ε, σχέσει του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να κάνουμε και τι σχετικές προσαρμογέ, προτάσει για προσαρμογέ στη βασική μα στρατηγική. Κύρια συμπεράσματα αυτή τη αναθεώρηση είναι ότι περισσότερε από τι χώρε αυτέ παρουσιάζουν εμβάθυνση, αλλά όχι επαρκή αλλαγή στην κατεύθυνση των σχέσεων τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική που έχει προσδιοριστεί από το έγγραφό μας για τις στρατηγικές με τις σχέσεις, στις σχέση με τρίτες χώρες δεν έχει αλλάξει και παραμένει το κύριο, ο κύριος καθοδηγητής μας στα προγράμματα δράσεως. Πλην όμως δεν θα πρέπει και να λησμονήσουμε ότι η εμβάθυνση των σχέσεων, ιδιαίτερως ε, μέσω της ανατολικής γειτονίας, εταιρική σχέση, συγγνώμη, θα αντικατοπτριστεί και στα ενδεικτικά προγράμματα η NPI και θα επανέλθω ε, λεπτομερέστερα στην ε, επισκόπηση της Ρωσίας και της Λευκορωσίας α αναφερθώ όμως πρώτα στο πλαίσιο αυτής της ενδιάμεσης αναθεώρησης μέσα από την ε, κρίση, την οικονομική ε, που ε, οδήγησαν σε, σε εξελίξει τη σχέση μας. Η ανατολική λοιπόν εταιρική σχέση στηρίζεται σε ένα όραμα για την εξέλιξη των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αρμενία, την, το Αζερβαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, τη Γεωργία και με πολλές συνόδους κορυφής κυρίως πέρυσι είδαμε πολλές αλλαγές τις οποίες καταγράφει υποχρεωτικά η ενδιάμεση αναθεώρηση, επισκόπηση. Κύριο στόχο εταιρική σχέση είναι να προσδιοριστούν οι όροι εκείνοι οι οποίοι θα επιταχύνουν την πολιτική σύνδεση και την οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και των, ανατολικών, των κρατών τη Ανατολική Γειτονίας και οι σχετικέ συμφωνίε σύνδεση με την εμβάθυνση ταυτόχρονα και των ε, την ανάπτυξη των χώρων ελεύθερων συναλλαγών και των συνθήκων ή συμφωνιών διευκόλυνση θεωρήσεων διαβατηρίων με βάση και τι προποθέσει που προσδιορίζουμε για τι σχέσει αυτέ, είναι οι κύριοι παράγοντε που καθοδηγούν αυτή τη διαδικασία και χρειαζόμαστε τη συνεχιζόμενη επαφή και και ε, διαπραγμάτευση με τις χώρες αυτές για να αναπτυχθούν περαιτέρω αυτές οι συμφωνίες. Η ανταπόκριση λοιπόν του NPI στην ανατολική εταιρική σχέση. Καλύτερα τι ανταπόκριση δόθηκε στο NPI. Θα θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένο. Στο Μάρτιο του 2009 χορηγήθηκαν πλέον 350 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη της ανατολικής εταιρικής σχέσης μέσω του NPI σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αναπτύχθηκαν τα σχετικά προγράμματα με τα ε, κονδύλια τα οποία στόχο έχουν την ανάπτυξη των, ε, θεσμικών, ε, των, των θεσμών εν γέννη, την περιφερειακή, και περιφερειακή συνεργασία και όσον αφορά την ανάπτυξη των, την οικοδόμηση θεσμών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει την ανάλυση των αναγκών ε, που υπάρχουν σε θεσμούς οι οποίοι χρειάζονται για να ολοκληρωθούν και να υλοποιηθούν υποχρεώσει που προκύπτουν από το νομικό αυτό πλαίσιο, ότι τα προγράμματα περιφερειακή ανάπτυξη που στηρίζονται και στην πολιτική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινούν να, λειτουργούν από το 2012. Η χρηματοδότηση τη πολυμερού διάσταση ανατολική εταιρική σχέση συνεπάγεται ταυτόχρονα και πολυθεματικέ πλατφόρμε με προγράμματα εργασία, τι λεγόμενε φλάξιμ, πρωτοβουλίε φλάξιμ, και τις σχετικές πρωτοβουλίες που περιμένουμε ότι θα δώσουν τελικά, σε μια, ε, θα δώσουν τελικά ως αποτέλεσμα μια γενική πολιτική και στάση απέναντι στον Νότιο Κάφκασο και την ανάπτυξη του Ανατολικού Euronest ως θετική συμβολή σε αυτήν την εταιρική σχέση. Επιπλέον αυτού του πολιτικού πλαισίου προσφέρει το, η Ανατολική Εταιρική Σχέση. Τα προγράμματα η NPI προσφέρουν και, προ, δυνατότητες για προσφορά στήριξης σε περιφερειακές πρωτοβουλίες συνεργασίας όπως τις συνεργασίες επί το Μαύρη Θάλασσας και, τη Βόρεια Διάσταση. Και επίσης θέλω να φερθώ πολύ όμω στην οικονομική κρίση η οποία ε, έπληξε βαρύτατα την περιοχή με διαφορετικές εκδηλώσεις ανά χώρα κάθε φορά που όμως ε, έδειξε και προβλήματα στα ισοσύγεια πληρωμών και προβλήματα ως προς το, στα ελλείμματα των προϋπολογισμών και ε, σημαντικά προβλήματα κόμματα προς την ανάπτυξη πολλών από τις χώρες αυτές. Στα πληρωμών και τα εθνικά ελλείμματα προτείνουμε περισσότερο μακροοικονομικές λύσεις σε συνεργασία με το Διεθνές Ρωσματικό Ταμείο και τα σχετικά πακέτα. Για τη Γεωργία και την Αρμενία ήδη έχουν κατευθεί σχετικές προτάσεις και θα επικεντρωθούμε ακόμη περισσότερο στους επενδυτικές μεθόδους και την ε, προαγωγή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των επενδυτικών διευκολύνσεων, όπως ονομάζονται, των οποίων ε, η πρικοδότηση θα ενισχυθεί σημαντικά, μαζί με την ε, δανειοδότηση του ENPI που θα ενισχυθεί επιπλέον. Το ENP και το ENB και η NBI θα επικεντρωθούν στο είναι ανακεφαλαίωση κυρίω για τις σημαντικέ τράπεζες και στην άμεση αναθεώρηση κατέστη επισαφέ ότι τα ENPI δεν μπορούν μόνο να αποτελέσουν βραχή πρόθεσμο μέσο. Μπορούν ωστόσο και πρόκειται να υποστηρίξουν την αηφόρο ανάπτυξη και την ανάκαμψη ε, στην περιφέρεια, υποστηρίζοντας μεταρρυθμίσεις και προσέγγιση προς τις προδιαγραφές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον και ε, το εμπόριο ή οι μεταφορές. Αν κοιτάξουμε τους τομείς προτεραιότητας της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των σχετικών κρατών, η χρηστή διακυβέρνηση, το PCA και τα, η εφαρμογή των προγραμμάτων δράσεων και οι κύριοι τομείς εταιρικής σχέσης, ε, κινητικότητα, ε, ενέργεια, επιχειρησιακό περιβάλλον, επιχειρηματικό περιβάλλον είναι τομεί που θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται και σε πολλές περιπτώσεις η στήριξη από τα ENPI αποτελεί και διατήρηση ή συντήρηση προηγουμένων προγραμμάτων. Θα ήθελα επίση να πω μερικά λόγια ως προς τις ιδιαιτερότητες του καθενός από τα κράτη αυτά. Για την Ουκρανία καταρχάς, με την οποία έχουμε, ε, η οποία είναι πρωταγωνιστεί στην Ανατολική Εταιρική Σχέση. Ακόμα δεν έχουμε δει τα αποτελέσματα των εκλογών, όμω και οι δύο υποψήφοι έχουν δεσμευτεί σε μια ατζέντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία θα συνεχίσουν να εστιάζονται με βάση την ε, οικονομική στήριξη ε, και τη Συμφωνία Σύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας, σχετική ατζέντα, το πρόγραμμα δράσεω και τη Συμφωνία Βίζα και ε, Επανισδοχή. Και το σχετικό πρόγραμμα θα επικεντρωθεί και στους οικονομικούς όρους, τη διαφάνεια που χρειάζεται, έτσι ώστε να προσελκυστούν ε, οι ε, επενδυτές που θα βοηθήσουν στην εξασφάλιση περισσότερων πόρων και αποδοτικότητας και περισσότερων εθνικών εσόδων. Ο τομέας της ενέργειας ε, είδε περισσότερη συνεργασία στο τομέα της μεταρρύθμισης του φυσικού, αερίου και μας απασχολεί ακόμη η Ουκρανία ως προς τον τομέα της, έρευνα, της ε, ενέργειας συγγνώμη, και της αποτελεσματικότητας ενέργειας. Η Μολδαβία τώρα, είναι εκ της κυβέρνηση έχει προευρωπαϊκές θέσεις και πρόγραμμα και παρουσιάζει, παρέχει ξέρετε ευκαιρίες για ε, προοδευτικές ε, μεταρρυθμίσεις και γι' αυτό ανταποκριθήκαμε και στο αίτημά για συμβούλους σε κύρια Υπουργεία. Θα αποστείλουμε λοιπόν συμβούλου και είναι η χώρα η πιο φτωχή από όλε τι ε, ανατολικέ εταιρικέ σχέσει που θα τη στηρίξουμε και όσον αφορά τα σχολεία και ε, άλλα μέσα που χρειάζονται ε, όπω επίση και σε μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη σχέση με την υπερδυστερία. Η Νότια Οσετία και η Αφχασία δεν είδαν να συνεχίζονται οι επαφέ μετά την κρίση του Οκτωβρίου του 2009, μετά τι προσπάθειε για την αποκατάσταση της ε, ομαλότητας. Ε, προσπαθήσαμε φυσικά πρώτα να αποκαταστήσουμε ε, τα προβλήματα που προκαλούν οι ένοπλες συγκρούσεις, να απαλύνουμε τον ανθρώπινο πόνο, να εξασφαλίσουμε τον επαναπατρισμό των εκτοπιστέντων και θα συνεχίσουμε με τα μέτρα ανάπτυξης εμπιστοσύνη επιπλέον τη υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη ελευθεροτυπία, τη ανάπτυξη κοινωνία των πολιτών, που είναι αντικείμενο του προγράμματο ΕΝΠΗ για την Γεωργία. Η υποστήριξη για την Αρμενία σημαίνει ιδιαίτερη έμφαση στο εμπόριο και την κανονιστική ε, σύγκληση εν ώψη της προετοιμασίας του ΕΝΠΗ και νέα ε, εστίαση σε ζητήματα κινητικότητας. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων συμβούλων ε, που παρακολουθεί την υπόθεση και την ε, εφαρμογή του προγράμματος δράσης του 2008, παρέχει και τις συμβουλές στην κυβέρνηση ως προς τους κύριους τομείς εφαρμογής του προγράμματος ΕΝΠΗ και του προγράμματος δράσης και ιδιαίτερα υποστηρίζει ε, και προσφέρει την αρρωγή της σε θέματα εξομάλυνσης ε, των αρμενοτουρκικών σχέσεων που βεβαίως θα στηριχθούν και οικονομικά από το ΕΝΠΗ. Ε, για το Αζερβαϊτζάν και το σχετικό πρόγραμμα δράσης ε, έχουμε βραδία πρόοδο. Ε, ανησυχητικά είναι τα θέματα της ελευθεροτυπίας, της ελευθερίας των μαζικής ενημέρωσης, της κοινωνίας των πολιτών, της ε, ελευθερίας του λόγου, όπου χρειάζεται επιπλέον υποστήριξη. Όσον αφορά την ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης του Ναγκόρνο Καραμπάχ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεθειμένη να προσφέρει εξειδικευμένη αρρωγή σε σχέση με κάθε πτυχή της ε, διευθέτησης των διαφορών και την ενίσχυση των σχετικών ε, παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών. Λευκορωσία, στη Λευκορωσία μεσοπρόθεσμη έκθεση καθυστέρηση για ένα χρόνο έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη και τα ε, συμπεράσματα του Συμβουλίου του περασμένου Νοεμβρίου για την εφαρμογή του ενδιάμεσου προγράμματος δράσης. Η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση θα λάβει υπόψη και τις πρόσφατες εξελίξεις των εκδημοκρατισμών, των ανθρωπινών δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου. Η, ε, το τωρινό ενδεικτικό πρόγραμμα, εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα θα παραταθεί κατά ένα χρόνο της να φτάσει μέχρι το 2011 η ε, διάρκεια του και μετά το καινούριο θα καλύπτει τα 2012 και 2013. Εν τέλει, συμπληρωματικές χρηματοδοτικές δραστηριότητε που θα περιλαμβάνουν και τη Ρωσία προέρχονται από περιφερειακά και διαπεριφερειακά κονδύλια του ENPI. Έχουν, προ... έχουν υποβαθμιστεί σιγά σιγά τα διμερεί προγράμματα, διότι η, Τουρκία, η Ρωσία δεν, έχει, δεν θέλει ούτε και χρειάζεται διμερή δράση. Απλώς στη διαπεριφερειακή συνεργασία με τα κρατη όπου η Ρωσία προσφέρει την, σε μεγάλο βαθμό τη χρηματοδότηση, τη βλέπουμε και τη δέσμευσή τη και σε τέτοια προγράμματα έχουμε ω τομεί και την ανώτατη εκπαίδευση και τα προγράμματα ανταλλαγών ε, ε, φοιτητών και τα λοιπά και την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Για να κλείσω, η υποστήριξη προσφέρει το NPI διδραματίζει σημαντικό ρόλο για τις προσπάθειές μας για ενίσχυση των ε, σχέσεων με τους εταίρους της ανατολικής ε, γειτονίας και ελπίζω ότι να μπόρεσα να περιγράψω τον τρόπο με τον οποίο το ENPI προσπαθεί να ενισχύσει την πολιτική συνεργασία, τη σύνδεση και την οικονομική ολοκλήρωση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαστε στη για κάθε ερώτηση και εγώ και οι συνάδελφοι ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Thank you very much. Ε, I have on my list Mr. Ευχαριστώ. Παρακαλώ κύριε με έχετε το λόγο. Σύντομα, Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση. Ελπίζουμε η συνέλευση της Euronest να συσταθεί στα τέλη Μαρτίου και να έχουμε αυτή την πολιτική πλατφόρμα για να συζητήσουμε όλα τα θέματα όπου θα υπάρχει και ανάμειξη όλων των εταίρων μας. Μία ερώτηση η οποία ίσως να θεωρηθεί κάπως προκλητική, αλλά φαίνεται πως για ορισμένους από τους εταίρους έχει δοθεί εντύπωση πως η προσθέμενη αξία αυτής της ε, εταιρικής σχέσης είναι το να γίνονται περισσότερες συνεδριάσεις ε, και σε ό,τι φορά τη χρηματοδότηση των ε, σχεδίων μάλλον προσδοκούσαν περισσότερα ναι, είναι μια νέα πολιτική, κονδύλια τα οποία έχουν ε, δοθεί σε αυτήν την ε, πρωτοβουλία είναι κάτι το καινούριο και για τα κράτη-μέλη αλλά και για τους ανατολικούς εταίρους και για την Κομισιόν φυσικά. Πώς αξιολογείτε τα προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί στο πλαίσιο αυτής της εταιρικής σχέσης και στο μέλλον στο εγγύς μέλλον προβλέπεται αύξηση των πόρων που χορηγούνται σε αυτές τις δραστηριότητε ε, ε, της Ανατολικής Σχέσης και μια ερώτηση σχετικά με τη Λευκορωσία. Δεν έχουμε συμφωνία συνεργασίας ε, ενδιάμεση συμφωνία δεν εφαρμόζεται, αλλά συμμετέχει στην ανατολική εταιρική σχέση η Λευκορωσία. Και έχει δείξει το ενδιαφέρον της για συμμετοχή και για άμεση ανάμειξη. Ο κ. Μινιγγέλη πρόσφατα στην επίσκεψή του είπε πως ε, προβλέπει να ξεκινήσει νέες διαδικασίες, νέες συζητήσεις. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα. Πιστεύει ότι θα υπάρξει ένα νέος πολιτικός διάλογος με τη Λευκορωσία μετά από το συμπέρασμα του Συμβουλίου πέρυσι. Ποια είναι η στρατηγική λοιπόν απέναντι στην Λευκορωσία. Αυτό είναι ένα ζήτημα που μπορεί να προκαλέσει κάποια προβλήματα σε εμά ε, σε συνδυασμό με την ε, σύσταση της ε, συνελεύσης γύρω Η κυρία Νέιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ και να ευχαριστήσω καταρχάς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση αυτή και την ανακοίνωσή της. Θα ήθελα να ρωτήσω αναφορικά με την κοινωνία των πολιτών σε όλες τις χώρες που συζητήθηκαν. Υπάρχει φιλοδοξία τουλάχιστον να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών στην εξέλιξη και την ανάπτυξη των προγραμμάτων, των ενδεικτικών προγραμμάτων, αλλά σε κάποιες χώρες δεν είναι εύκολο αυτό λόγω της γενικότερης κατάστασης. Θα ήθελα λοιπόν να μας διευκρινίσετε πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα αυτό. Άλλες ερωτήσεις από άλλους συναδέλφους. Ο κύριος Κιν. Για να απαντήσει εκτός μικροφώνου. I, um, Νομίζω ότι κοιτώντας την ε, ανατολική εταιρική σχέση, η οποία ασφαλώς ε, βρίσκεται σε φάση ε, εκτέλεσης, υπάρχει μια διμερής διάσταση και νομίζω ότι έχουμε σαφείς στόχους για το τι προσφέρουμε στους εταίρους μας. σύναψη μία συμφωνία εταιρική σχέσης εφόσον πληρούνται οι όροι συμπεριλαμβανομένης μίας ε, εμπορικής ε, συμφωνίας η οποία θα διευκολύνει την κινητικότητα των πολιτών και θα ενισχύσει την συνεργασία σε διαφόρους τομείς όπως στην ενέργεια. Νομίζω ότι είναι σαφές το τι προσφέρεται και η δική μου εντύπωση είναι ότι ήταν θετική η ανταπόκριση εκ μέρους των εταίρων μας. Όπως είπατε και εσείς, Πρόεδρε, στην εισαγωγή σας, βρισκόμαστε σε φάση διαπραγμάτευσης ε, συμφωνιών εταιρική σχέσης με δύο χώρες, με την Ουκρανία και την Μολδαβία και προετοιμάζουμε οδηγίες διαπραγμάτευσης στο στο εσωτερικό του Συμβουλίου για τα τρία κράτη του Καυκάσου. Σε ό,τι αφορά την πολυμερή διάσταση τώρα, νομίζω ότι ένα από, από τα καινοτομικά στοιχεία της ανατολικής συντερικής σχέσης είναι ακριβώς το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η πολυμερή διάσταση, η οποία θεωρώ ότι θα προσελκύσει και θα ομαδοποιήσει τους εταίρους μας για τον περαιτέρω διάλογο. προκειμένου να κατανοήσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές, το ευρωπαϊκό και εκτιμένο σε διάφορους τομείς. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα καινοτομικό στοιχείο το οποίο υποτέχθηκαν με ενθουσιασμό όλες οι χώρες. Σε ό,τι αφορά τα κονδύλια, δεν κατάλαβα ακριβώς την ερώτηση αυτό που αναφέρουμε για τα ενδεικτικά προγράμματα είναι η περίοδος 2011 με 2013. Σε ό,τι αφορά την, τα κονδύλια των 50 εκατομμυρίων ευρώ, θα αρχίσουμε ήδη το 2010 να εκτελούμε προγράμματα και θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα αν θα υπάρξουν επιπλέον πόροι. Αυτό προφανώς θα εξαρτηθεί και από τον προϋπολογισμό και από την διαθεσιμότητα κονδυλίων. Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε. Γιατί Λευκορωσία, να πω το εξής. Όπως ξέρετε, το 2008 διατυπώσαμε τους πέντε τομείς όπου θα θέλαμε να σημειωθεί πρόοδος προκειμένου να έχουμε πιο εντατικές σχέσεις με τη Λευκορωσία. Αναστολή της ε, απαγόρευσης ε, των θεωρήσεων και το Συμβούλιο ζήτησε την εφαρμογή δύο ενεργειών. Καταρχάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτιμάσει μια πρόταση για το κοινό ενδιάμεσο σχέδιο, το οποίο αποτελεί, αν θέλετε, ένα σκιώδες σχέδιο δράσης, ελήψη μιας πιο σημαντική σχέσης με την Λευκορωσία και δραστηριοποιούμαστε λοιπόν στο μέτωπο αυτό και επίσης το Συμβούλιο ζήτησε να προετοιμαστούν οδηγίες διαπραγμάτευσης εφόσον ευνοήσουν και οι πολιτικές ε, συνθήκες να ξεκινήσουν ε, οι διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες για θεωρή και για τις συμφωνίες επανεισδοχής. Προσπαθούμε λοιπόν να ενθαρρύνουμε την πρόοδο στους πέντε τομούς, τομείς αυτούς και ενημερώνουμε τις αρχές για το τι θα επιτευχθεί και τι τους προσφέρουμε αν επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση που κάνατε για την κοινωνία των πολιτών, γενικά πρέπει να πω ότι έχουμε πολλές επαφές με την κοινωνία των πολιτών. Στο πλαίσιο της κατάρτισης ε, των εκθέσεων πρόοδου, εκθέσεων βάση των ε, εμπειριών και των πληροφοριών που δεχόμαστε από την κοινωνία των πολιτών. Προσπαθούμε επίσης να διαβουλευτούμε με την κοινωνία των πολιτών σε ό,τι αφορά τα σχέδια δράσης τα σχετικά. Thank you. Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ επίση για τι εξήγησει που είδαμε μέχρι τώρα. Ξέρετε ότι καταρχά η πολιτική αυτή την χάνει τη υποστήριξη του Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή μα, ιδιαίτερα όσο έχουμε κάθε πολιτικό συμφέρον στη σχέση με τα κράτη αυτά, να προοδεύσουμε. Ερώτησή μου λοιπόν οι οποίε θα μπορούσαν να επιτρέψουν να δούμε με πιο συγκεκριμένο μάτι τι πολιτικέ αυτέ και τι σχέσει με τα κράτη αυτά. Θα ήθελα να μα πείτε για το κάθε κράτο ένα συγκεκριμένο σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το οποίο αισθάνεστε ιδιαίτερα υπερήφανο. Για να δούμε τι σημαίνει αποτελεσματικότητα, τι σημαίνει εύστοχη πολιτική, τι σημαίνει επιτυχία αυτών των σχεδίων. Για να μπορούμε να πούμε και στους πολίτες μας ότι τα χρήματά τους πιάνουν τόπο. Ε, για την Αρμενία, για το Αζερβαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία. Ένα παράδειγμα μπορείτε να μας δώσετε. Κάναμε αυτό, το σχεδιάσαμε από το 2007 και τώρα το 2010 ε, βλέπουμε ότι έχει τα εξής καλά αποτελέσματα. Κάτι που μπορώ και εγώ να το σημειώσω και να πάω μετά στους ε, συμπατριώτες μου, στους ψηφοφόρους μου και να τους πω να τι κάνουμε εμείς εκεί. κύριος Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θα σας ξεφνιάσετε ότι με απασχολεί το θέμα της Λευκορωσίας ιδιαίτερος. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ και στα όσα είπε ο κύριος Βεγγένιν και την ε, το έγγραφο, το οποίο είναι κατά πάσα πιθανότητα το μόνο έγγραφο που έχει δημοσιεύσει η Επιτροπή σε σχέση με, την Ευρωπαϊκή, με το Ευρωπαϊκό Μέσο Εταιρική Σχέση και Συνεργασία ε, που αφορά την ε, Λευκορωσία, γιατί αυτή η έκθεση δεν αφορά τη Λευκορωσία. Ίσως λοιπόν, ίσως θα μπορούσα τώρα να σας ρωτήσω, διότι στο δεύτερο τμήμα ε, της περίοδου αυτής της πενταετίας 2007-2013 στη φάση αυτή που βρισκόμαστε τώρα θα πρέπει να δούμε το επόμενο το δεύτερο κομμάτι δηλαδή αυτής της πενταετίας και έχουμε τους δύο μεγάλους πυλώνας για την άποψή μου πρέπει να υποστηρίξουμε καταρχάς να ε, εισαγάγουμε και να ολοκληρώσουμε την ε, συμφωνία για τη διευκόλυνση θεωρήσεων διαβατηρίων έτσι ώστε να βοηθήσουμε στους ανθρώπους αυτούς να αναπτύξουν τις σχέσεις τους κινητικότητα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τη Λευκορωσία. Αλλά και ο δεύτερος πυλώνας είναι πολύ σημαντικός, εκ παραλλήλου δηλαδή με τις διαπραγματεύσεις με τις αρχές της Λευκορωσίας που προχωρούν ταχύτατα και ως είπε και ο συνάδελφος νωρίτερα ε, είναι και πολλά υποσχόμενες, σημειώνω ότι εκ παραλλήλου οι αρχές της Ρευκορωσίας είναι πολύ αυστηρές και προσπαθούν να περιορίσουν κάθε μορφή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν όταν κοιτάμε τα α, στοιχεία, τα αριθμητικά, τα σχετικά με τον προϋπολογισμό ε, που προβλέπεται για τη Λευκορωσία στο Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα, μόνο 20 εκατομμύρια και το δέχομαι βεβαίως διότι έχει ιδιαίτερες συνθήκες η Λευκορωσία, μόνο το 70% της Λευκορωσίας πήγαινε στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και το υπόλοιπο στην οικονομική στην κοινωνική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση. Το δεύτερο αυτό κομμάτι που είναι απολύτως απαραίτητο δεν θα πρέπει να έχει περισσότερα χρήματα ως πρικοδότηση υποστήριξη των δημοκρατικών εξελίξεων και της χρηστής διακυβέρνησης. Είναι απολύτω απαραίτητα αυτά για τη Λευκορωσία. Γιατί οι αρχέ τη Λευκορωσία, όπω είπα, κάνουν ό,τι μπορούν για να θέσουν εκτό παιδιά ή εκτό δράσης την κοινωνία των πολιτών και κάθε άλλο εκπρόσωπο των πολιτών, ακόμη και τι οργανώσει που είναι πολύ μετριοπαθεί και που ακολουθούν ή επιδιώκουν μια σταδιακή διαδικασία εκδημοκρατισμού. Η κυβέρνηση προσπαθεί να τους πέταξει όλους έξω λοιπόν, να τους αποφύγει, να τους θέσει στο περιθώριο. Κάθε μορφή αντίδρασης ή αντιπολίτευσης που θα μπορούσε να συμμετέχει σε σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκορωσίας και βέβαια προσπαθεί να την θέσει εκτός παιδιάς. Άλλες ερωτήσεις λέει ο Πρόεδρος. Καλώς ο κύριος και για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ και θα απαντήσω στην τελευταία ερώτηση καταρχάς. Για να μετά από τον συνάδελφο τον Διευθυντή Κανάρη να δώσει κάποιες απαντήσεις στα υπόλοιπα ερωτήματα. Και η προτασία της ξέρουμε ότι ενδιαφέρει πολύ η Λευκορωσία και, έχετε και έχουμε πάντα πολύ καλή συνεργασία μαζί σα και σχέσεις. Ε, θα ήθελα να πω ότι ως προς την αδιευκρίνηστη ακόμη πολιτική κατάσταση ε, που παρατηρείται ε, ήταν αυτή και ο λόγος για τον οποίο ε, χρειάστηκε να προσθέσουμε ένα χρόνο ακόμα ή να καθυστερήσουμε κατά ένα χρόνο ακόμα το πρόγραμμα. Τα στοιχεία που βλέπετε λοιπόν είναι ακόμη πιο προσωρινά γιατί μένει ακόμα ένας χρόνος για να ολοκληρωθεί αυτή η φάση. Άρα ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μία ε, δυνατότητα να ε, καλύψουμε τα κενά ενδεχομένως με την ε, διάμεση αναθεώρηση που θα γίνει σε ένα χρόνο. Επίσης θέλω να σημειώσω ότι αυτά τα οποία συζητούμε εδώ προφανώς είναι οι δυνατότητες στήριξης από το ENPI μέσω των εθνικών ενδεικτικών προγραμμάτων. Υπάρχουν και άλλοι μέσα συνεργασίες όπως η ε, ενίσχυση σχετική με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνία των πολιτών που αναφέρατε και εσεί, σε παραδείγμα το μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ή επί παραδείγματι το μέσο που ονομάζεται μη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές, δηλαδή μέσα τα οποία προσφέρουν χορηγίες μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και συγκεκριμένους στόχους για την περιοχή και πιστεύω ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία και αποτελεσματικότητα για την ε, Λευκορωσία. από τη Europe, πρόεδρε, να μου επιτρέπετε να δώσω κάποιε στοιχεία προς την εφαρμογή των προγραμμάτων στην γειτονία. Και θα ήθελα να σημειώσω ότι πολύ ευχαριστώ να διαθέσω και τι αιτήσει εκθέσει μα που δίνουν ακόμη πιο λεπτομερεί συμπεράσματα και αποτελέσματα των εργασιών μα στον κύριο Βουλευτή. Αλλά να δώσω κάποια πρόχειρα παραδείγματα, ότι, ότι εγώ δηλαδή χρησιμοποιώ ω παράδειγμα για να εξηγήσω την πολιτική γειτονία. Ε, εκ του προχείρου λοιπόν από τη σημερινή ακόμη διάσκεψη για τις παγωμένες ε, στον πάγο ε, συγκρούσεις Έχουμε χρηματοδοτήσει επί ένα χρόνο τουλάχιστον για τη Μολδαβία ε, την ε, υποστήριξη των αστυνομικών θεσμών ε, και δομών αλλά και των τελωνιακών αρχών κατά τρόπον ολοκληρωμένο με συμμετοχή και πολλών από τα κράτη-μέλη και ταυτόχρονα όχι μόνο αναφερόμενοι μόνο στην Μολδαβία αλλά και στην άλλη πλευρά των συνόρων και τα, στην περιοχή περί την υπερθυνιστερή έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, περιορίσουμε τις δυσάρεστες ή τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί βεβαίως η διαφθορά, το μέζο το, ε, και το διεθνές έγκλημα σε μια περιοχή με ε, τέτοιου είδους συγκρούσεις αλλά ταυτόχρονα και στα θέματα των τελωνίων ε, ή των συνοριακών ελέγχων ε, βλέπουμε ότι για την υπερδυνιστερία την ίδια μπορούμε να έχουμε σωστικά αποτελέσματα ή για τη δικαιοσύνη στην Ουκρανία και τη Μολδαβία στην Ουκρανία μπορέσαμε παραδείγματι να έχουμε ακόμη πιο στενές σχέσεις ε, και να συνδυάσουμε την βοήθεια προσφέρουμε ως προς την υποχρέωση ε, για επανεισδοχή. Για τη Γεωργία νομίζω πιο εντυπωσιακές προσπάθειες και με πολύ καλή ε, υποστήριξη και από εσάς ήταν η προσπάθεια για στήριξη των εκτοπιστέντων. Μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ως προς το φρονιστικό σύστημα που αφορούσε τους ανουλίκους που ήταν πραγματικά συγκλονιστικοί Είχε πάρα πολύ κακέ συνθήκε τόσο για την ποινική διαδικασία όσο και για τι συνθήκε κράτηση. Δηλαδή και συνθήκε στη δίκη, αλλά και συνθήκε κράτηση στα ιδρύματα ανηλίκων. Ε, εκεί βλέπουμε πολλά θετικά, πολλές θετικές εξελίξεις. Ένα πολύ δύσκολο θέμα οφείλω να ομολογήσω. Για τη δε Αρμενία έχουμε μπορέσει την ε, επαγγελματική κατάρτιση να την θέσουμε ως στην πρώτη γραμμή του συστήματος ε, του εκπαιδευτικού για το Αζερβαϊτζάν ιδιαίτερα στην ε, αποτελεσματικότητα της ενέργειας έχουμε δώσει έμφαση και κοιτάμε την ενεργειακή την αποτελεσματικότητα της ενέργειας όχι μόνο στα ε, νοικοκυριά αλλά και ως προς την ε, καύση, δηλαδή ως προς την ε, ρήπανση του περιβάλλοντος κτλ. Σε όλα αυτά βλέπουμε ουσιαστικά αποτελέσματα από το Αζερβαϊτζάν ήδη πέρυσι ολοκληρώθηκαν 6-7 συμβάσεις που επιτρέπουν και την εμπλοκή μιας νεοεμφανιζόμενης θα έλεγα κοινωνία των πολιτών καλά αποτελέσματα είναι αυτά, καλά παραδείγματα είναι αυτά. Είναι εκεί που έχουμε δείξει ότι μπορούμε να καθοδηγούμε και όλα στην πολιτική επικαιρότητα και να αποδεικνύουμε ουσιαστικές επιτυχίες. Πρόεδρε, να προσθέσω δύο δράσει οι οποίε καταδεικνύουν νομίζω με καλό τρόπο ότι προσπαθούμε να πετύχουμε. Καταρχά, μία ομάδα υψηλά βαθμών συμβούλων, οι οποίοι στην οποία αναφέρθηκα και στην εισαγωγή μου, την οποία αποστήλαμε στην Αρμενία. Και ακριβώς αυτή είναι η αντίδραση στις ανάγκες της Αρμενίας σήμερα, προκειμένου να βοηθήσουμε την ε, κυβέρνηση να εντοπίσει τα ζητήματα ως προς την οικονομική ενσωμάτωση στα πλαίσια της ε, ανατολικής Τερικής σχέσης να εντοπίσει τις ανάγκες της λοιπόν. Και αυτό το εκτιμούν ιδιαίτερα οι αρχές της Αρμενίας. Και να πω ότι αυτό το κάνουμε ανταποκρινόμενοι στην ε, νέα κυβέρνηση. Στο τέλη Ιουλίου αποστήλαμε δύο οικονομικούς συμβόλους και τώρα αποστέλουμε μια πιο Μεγάλη ομάδα. Επίσης για τη Γεωργία. Να πω ότι υποστηρίζουμε εν μέρη, μάλλον ε, η χρηματοδότηση είναι εν μέρη από την Ανατολική Τερική Σχέση και, και εν μέρη από το μέσο σταθερότητας. Και καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των εσωτερικών εκτοπιστέντων μετά το 2008. Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη δυναμικού στην ε, τοπική κοινωνία των πολιτών. Υποστηρίζουμε θέματα διατησίας και παρέχουμε γενικότερη υποστήριξη στο πλαίσιο αυτό. Αυτά νομίζω ότι αποτελούν συγκεκριμένα μέτρα που είναι πολύ ωφέλιμα. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κανεί άλλο το λόγο. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ολοκλώσουμε τι εργασίε μα. Σα υπενθυμίζω πω στι 6 θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με την Μάρντεν Ολμπράιτ και του συνεργάτε τη σχετικά με την αναθεώρηση τη στρατηγική αντίληψη για τον ΝΑΤΟ. 18 και 30 σε 25 λεπτά, 27 για την ακρίβεια. Ευχαριστώ. Γεια σας.